Good morning, colleagues. If there are no objections to the agenda, it is adopted. Συνάδελφοι, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται. Να σας πω επίσης ότι δεν έχουμε κροατικά σήμερα, μαλτέζικα και γουαντελικά. Κροατικά, μαλτέζικα και τελικά δεν θα υπάρχουν ούτε αύριο. Να εγκρίνουμε τις συστάσεις των συντονιστών. Σύμφωνα με τον άρθρο 205 έχουμε τον διορισμό των εισηγητών. Η κυρία και από τους Σοσιαλδημοκράτες διορίστηκε για την ε, έκθεση ίδια ε, πρωτοβουλία για τη στρατηγική με την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική. Εγκρίθηκαν λοιπόν οι σχετικέ συστάσει. Εγκρίνονται ηλεκτρονική ψηφοφορία στι 12 σήμερα για τι ε, συνθήκε τη φυλακή. Και αν Είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε στο σημείο 3 της ημερησίας διαταξής μας. Συνάδελφοι, σήμερα έχουμε τον κύριο Άντρη Σέιτσελ μαζί μας, ε, επικεφαλές της Μόνιμης Επιτροπής για την Ασφάλεια. Η σημερινή παρουσίαση θα εστιαστεί στη σημαντική εργασία που έχει γίνει από την Επιτροπή τους τελευταίους έξι μήνες, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα αναφέρει ο καλεσμένος μας. Καταρχάς, στις 21 Απριλίου η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έλαβε μια παρουσίαση σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα και την αξιολόγηση των απειλών και σε ό,τι αφορά τον κύκλο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018 με 2021, όπου συγκεκριμένοι στόχοι και στρατηγικές ερμηνεύοντας μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήμου. Και στη συνέχεια, στις 18 Μαΐου, η Σχετική Επιτροπή ενέκρινε τι νέε προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τα επόμενα χρόνια. Άρα προσβλέπουμε στην παρουσίασή για τα θέματα αυτά. Κατά δεύτερα, το θέμα των συστημάτων ε, των πληροφορικής και της δια λειτουργικότητα. Η Επιτροπή Τζουλιά Κίνγκ παρουσίασε στι 29 Μαΐου την τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου για τα συστήματα ενημέρωσης και τη διαλειτουργικότητα. Ακούσαμε λοιπόν το συντονιστή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τον επικεφαλής για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τον επιβλέποντα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σήμερα λοιπόν μπορούμε να ακούσουμε και την παρέμβαση της ΚΟΖΗ για το σημαντικό αυτό θέμα. Κύριε Σέιτσελα, έχετε το λόγο για να μας κάνετε τη σημαντική αυτή παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σαφή αυτή εισαγωγή σας. Καλημέρα αξιότιμοι βουλευτές κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη, μεγάλη τιμή να σας ενημερώνω ως πρόεδρος της ε, μόνιμης ε, συνεργασίας για την εσωτερική ασφάλεια. σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τη Επιτροπή. Οι τελευταίοι έξι μήνε ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντε. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η περίοδο για τη χώρα μου και για μένα προσωπικά και πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι έγινε σημαντική πρόοδο σε διάφορα σημαντικά ζητήματα, όπω τα γνωρίζετε. Η κόζη συναποκαλείται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των κρατών μελών και γενικούς διευθυντές ε, σε επίπεδο προσωπικού που είναι αρμόδιοι για θέματα που άπτονται της ιστορικής ασφάλειας. Για τα συγκεκριμένα ζητήματα συμμετέχουν και εκπρόσωποι από τη Europol, τη Eurojust, τη Cipol, τη Frontex, την Αγιλίζα και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Στη σημερινή μου παρέμβαση θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα. Το πρώτο, αδελαγή πληροφοριών και διαλειτουργικότητα και ο κύκλος πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις πιο σημαντικές ε, δραστηριότητες της ΚΟΖΗ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας είναι να εξασφαλίσουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Και υπάρχουν δύο πτυχές σε ό,τι αφορά την εργασία της ε, ΚΟΖΗ. Καταρχάς, η ΚΟΖΗ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του οδικού χάρτη για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ άλλων και λύσεις διαλειτουργικότητας στον τομέα της δικαιοσύνη ε, και της εσωτερική ασφάλειας. Ε, αυτό εγκριθήκε από το Συμβουλίο πριν από ένα χρόνο υπό την Ολλανδική Προεδρία. Όπως ξέρετε, περιλαμβάνει αυτός ο οδικός χάρτης 50 δράσεις για να εξασφαλίσουμε ότι όλες ε, οι δράσεις συντονίζονται οι βάσεις δεδομένων ότι ενημερώνονται τακτικά και ότι επιτόπου οι παράγοντες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Υπό την Προεδρία μας ε, ε, προετοιμάσαμε τη δεύτερη εφαρμοστική έκδοση του δικού χάρτη. Εστιαστήκαμε στην αύξηση της συνταλλαγής ε, πληροφοριών και στη χρήση διαφόρων συστημάτων πληροφοριών. Για παράδειγμα, ο αριθμός των ετοιμάτων για το σύστημα της ε, Interpol διπλασιάστηκε και πλέον από το 2015 μέχρι το 2016. Μισό εκατομμύριο περίπου το 2015, 1,5 εκατομμύριο τίματα το 2016. Και η χρήση του συστήματος ε, ΣΥΣ επίσης αυξάνεται. Και ο αριθμός ε, των ε, alerts έχει επίσης αυξηθεί. 60.000 το 2015, σημάνσεις το 2015. Και φέτος είμαστε ήδη πάνω από 106.000 ε, σημάνσεις. Συνεχίζονται επίσης να αναπτύσσονται οι συνδέσεις, οι λειτουργικές συνδέσεις και υπάρχουν 23 κράτη-μέλη στην παρούσα φάση που συνδέονται για την ανταλλαγή δεδομένων DNA και άλλα 22 τα οποία συνδέονται για την ανταλλαγή τακτικών αποτιμωμάτων και στοιχείων για δικά οχήματα. Το 2016 τα κράτη-μέλη αύξησαν τη χρήση των δεδομένων της Interpol για τα έγγραφα σε SLTD είναι γνωστή αυτή η βάση δεδομένων και οι ονομαστικές βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους τρομοκράτες μαχητές. Και αυτή η τάση παρατηρείται ότι συνεχίζεται το 2017 γιατί έχουν διπλασιαστεί τη χρήση των βάσεων δεδομένων αυτών από το 2015 μέχρι το 2016. Και επίσης ήταν πολύ πιο αυξημένες ε, το, τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017 σε σχέση με όλο το χρόνο του 2016. Δεύτερη Δεύτερο τομέα είναι η διαχείριση πληροφοριών σε ό,τι αφορά την εργασία τη ΚΟΖΗ για να υπάρχει διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφόρηση για την διαχείριση των συνόρων, των μεταναστευτικών ροών και τη ασφάλειας. Στην Προεδρία μας, λοιπόν, παρακολουθήσαμε στενά το θέμα αυτό του σύστημα αυτό των συστημάτων όπως το είχε καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επί της βάσης αυτής το συμβόλιο που συνέλθε στις 8 Ιουνίου καλωσόρισε τις συστάσεις της υπηρεσίας της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την επιτεύξη της ε, διαλειτουργικότητας και διάφορες αντιπροσωπείες τόνισαν ότι η πρόοδος σε αφορά θέματα διαλειτουργικότητας αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές τους. Μία από τις δεσμεύσεις του Συμβουλίου που παρουσιάζεται και στα πορίσματα αυτά είναι να συνεχίσει να παρακολουθεί τις συζητήσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου που έχει που παρακολουθούνται σε μια ειδική μορφή και επιτροπή του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου. Χθε λοιπόν η Κόζη, επί της βάσης αυτής, συζήτησε την πρόταση της ε, επερχόμενης Προεδρίας να συσταθούν διάφορες επιτροπές και διάφορες ε, συνθέσεις για να συζητηθούν τα θέματα διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων στο θέμα της δικαιοσύνης και των αστρικών υποθέσεων και ήδη έχουμε πετύχει σχετική συμφωνία. Και οι φίλοι της Προεδρίας θα εστιαστούν κυρίως σε τρία ζητήματα. Το πρώτο, να συζητηθεί το αποτέλεσμα των ε, μελετών εφικτότητας για διάφορα ζητήματα διαλειτουργικότητας. η τροφοδότηση των συστημάτων από την Κομισιόν και η ενημέρωση του δικού χάρτη και η συνέχιση της εφαρμογή του όπου αυτό χρειάζεται προκειμένου να είναι πραγματικά ένα ενιαίο εργαλείο στα πλαίσια του Συμβουλίου και να δοθεί έτσι σωστός τρόπος παρακολούθησης των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Αυτό θα γίνει υπό την ε, στρατηγική καθοδήγηση της ΚΟΖΗ για να μπορούμε να παρακολουθούμε στενά την, εξελίξει τις εξελίξεις ε, στον τομέα αυτό. Θα περάσω λοιπόν στον Ευρωπαϊκό Κύκλο Πολιτικής το 2017 ήταν ε, το πρώτο έτος ε, για τον νέο αυτοπολιτικό κύκλο και μπορούμε να πούμε ότι ο πολιτικός κύκλος 2014-2017 θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο φέτος. Ταυτόχρονα χρειάστηκε να ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες για το νέο κύκλο πολιτικής 2018-2021 για να επιλέξουμε σωστά το βασικό θέμα του επόμενου πολιτικού κύκλου, κυρίως διαλέξαμε τη μεθοδολογία για την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πρόοδων στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος, που βασίζεται στη συνεργασία μυστικών υπηρεσιών και που καλύπτει πολλούς κύκλους ετών. Οι προτεραιότητες μας εντοπίζονται βάσει των ε, μυστικών πληροφοριών που διαθέτουμε και της αξιολόγησης για το σοβαρό και διεθνές έγκλημα. Ίσως να το γνωρίζετε πιο καλά με τα αρχικά του. Ε, είναι η εκθέση ΣΟΚΤΑ που ε, συντάσσει η Europol. Η έγκριση αυτών των προτεραιοτήτων και του πολιτικού κύκλου σημαίνει ότι θα ξεκινήσει η υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων δράση στο νέο πλαίσιο του ονομαζόμενου νέου επιχειρησιακού κύκλου. Και στο τέλο του κύκλου αυτού θα διεξαχθεί και πάλι αξιολόγηση όπω πάντα. Σημαντικό επίση να πούμε ότι ω προ τον κύκλο 2014-2017 Η αξιολόγηση έγινε από ανεξάρτητο φορέα. Ο αξιολογητής απελέγει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι και τα απορίσματα της αξιολόγησης υποβλήθηκαν στην Κόζη φέτος το Φεβρουάριο. Τα απορίσματα αυτής της αξιολόγησης τα υποβάλαμε στην φάση προετοιμασίας ε, του νέου πολιτικού κύκλου που θα καλύπτει το 2018-2021 όπω είπα ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά, πιο δραστικά, ευθυγραμμισμένα και light, πιο light, πιο ελαφρά. Όταν λέω πιο ε, ελαφρά εννοώ λιγότερο άχθος, δηλαδή λιγότερη υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και περισσότερη έμφαση στις κινητρές δυνάμεις της κάθε προτεραιότητας που θα πρέπει αυτές κυρίως να συντάσσονται προσεκτικά. Μια άλλη αλλαγή είναι ότι από την ε, Europol θα υπάρχει σύνταξη από το 2019 η έκθεση ΑΜΕΤ που είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτικού κύκλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κρυθεί ήδη αν θα έχει πετύχει ο κύκλος ή όχι, απλώς Ελπίζουμε να είναι ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία του. Ε, θέλουμε να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα με συγκεκριμένε δράσει για να αντιμετωπίσουμε οργανωμένα δίκτυα, ε, να κατασχέσουμε περιουσιακά στοιχεία, παράνομα ε, εμπορεύματα ή ναρκωτικά και να εμποδίσουμε την εμπορία ανθρώπων καταπολεμώντα του διακινητέ μεταναστών. Λόγω χάρη κατά τι κοινέ ημέρε δράση το 2016 που είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Κύκλου Δράσης, 529.500 ε, αρχές συναντήθηκαν και συζήτησαν ότι τουλάχιστον 600 ύποπτοι συνελήφθησαν, 539 θύματα εμπορίας εντοπίστηκαν, 745 μετανάστες διασώθηκαν και κατασχέθηκαν 38 τόνοι κοκαίνης. Ο νέος πολιτικός κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 28, 27 και 28 Μαρτίου φέτος. Αυτό βεβαίως μας ικανοποίησε τα μάλλα. Πρώτο στοιχείο του πολιτικού κύκλου είναι η αξιολόγηση των απειλών. Στις 9 Μαρτίου φέτος η Europol εξέδωσε την αξιολόγηση απειλών σοβαρού εγκλήματος και οργανωμένου εγκλήματος, τη γνωστή και ως όκτα, η οποία έδειξε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5.000 ε, ομάδες ε, οργανωμένου εγκλήματος που δρούν σε διεθνές επίπεδο και αυτή τη στιγμή ερευνώνται με ανακριτικές δραστηριότητες όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ περίπλοκη διοργάνωση και με ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα. Η EU Όκτα, αυτή η έκθεση έχει γίνει βάση για τον εντοπισμό των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμηθεί το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Το δεύτερο βήμα του πολιτικού κύκλου. Συζητήσαμε τις συνιστόμενες ε, προτεραιότητες της ΟΚΤΑ σε πολλές συναντήσεις και λάβαμε υπόψη τα σχόλια των κρατών μελών των ε, φορέων τους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως την έκτη έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε στις 17 Ιουνίου. Οκτώ βασικές προτεραιότητες πρότανε η έκθεση 8, για να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρότερες απειλές σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Πέντε συγκεκριμένες προτεραιότητες για τις εγκληματικέ δραστηριότητες και τρεις που αφορούν περισσότερο από ένα τομείς. Οι τρεις συγκεκριμένες απειλές εγκλήματος, ήταν το κυβερνοέγκλημα, η παραγωγή ναρκωτικών, η, διάδοση, η εμπορία τους, οι οργανωμένες διαρρήξεις και κλοπές, κυρίως ε, οι κλοπές περιουσιακών στοιχείων και εμπορία ανθρώπων. Κυρίως μας ενδιέφερε το παράνομο κέρδος και η λεύκανση παράνομων προσόδων το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Επίσης τα παραποιημένα αγαθά και υπηρεσίε, Τα παράνομα αγαθά και υπηρεσίε. Με τις πετολιώτες αυτές δώσαμε έμφαση από την Προεδρία να επιλέξουμε και να δράσουμε σε κάποιες από αυτές για να βρεθούν πολιτικές λύσεις καθώς αυτό θα έχει και σοβαρό αντίκτυπο στους ανθρώπινους πόρους των κρατών μελών. Έχουμε εντοπίσει 10 δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του εγκλήματο. Ενώ στον προηγούμενο πολιτικό κύκλο είχαμε νέα. Για να τις αναφέρω. εγκλήμα, ναρκωτικά και ιδίω η κάναβη, η κοκαίνη, η ηρωίνη, τα συνθετικά κοινέ ψυχοτρόπε ουσίε. Προφανώ εδώ υπάρχει κάποια πιστοχώρηση στο νομικό επίπεδο. Οργανωμένο έγκλημα και τα περιουσιακά του στοιχεία. Διακίνηση ανθρώπων. Η απάτη και η φόρη πολυτελείας η παράνομη εμπορία αποβλήτων και η ανάκτηση περιοδικών στοιχείων από το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι περισσότερες από τις προτεραιότητες αυτές είναι απλώ η εξακολούθηση των προτεραιοτήτων που είχαν εντοπιστεί στον προηγούμενο πολιτικό κύκλο. Αυτό που βλέπουμε είναι το περιβαλλοντικό έγκλημα ως μια νέα προτεραιότητα. Κάτι που εντοπίστηκε ως μείζον απειλή στον προηγούμενο κύκλο μεταξύ των ε, κερδών και του ξεπλήματος ε, βρώμικου χρήματος. τα παραποιημένα αγαθά δεν θα είναι πλέον ε, ξεχωριστή προτεραιότητα. Θα εντάσσεται στην ε, στα έσοδα του οργανωμένου εγκλήματο. Κατόπιν αυτού, οι συζητήσει στην ΚΟΖΗ ασχολήθηκαν με το να εντοπίσουν, για τα κράτη, να αυτά τα κράτη-μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν. Για να επεξεργαστούμε στατικικούς στόχους και επιχειρησιακές δράσεις. Η διαδικασία κοντεύει να ολοκληρωθεί, αλλά συνεχίζεται. Τα συζητήσαμε διεξοδικά στην ε, συνάντησή μας και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα εμφανιστούν και άλλες χώρες που θα συμμετάσχουν και κάποιες έχουν ε, σκοπό να αναλάβουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτά θα συζητήσουμε τις ερχόμενες ημέρες και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα ήδη ως το τέλο της εβδομάδας. Επίσης να σας πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα στις 26 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώσει και θα εκδώσει μάλλον, ε, μάλλον θα οργανώσει ένα διαστήριο για το στρατηγικό πρόγραμμα αυτής της χρονιάς όπου θα ορίσει τους ελάχιστους οριζόντες στρατηγικούς στόχους για όλες τις, οργανω... τις προτεραιότητες μετά του οργανωμένου εγκλήματος στον ε, Ευρωπαϊκό Κύκλο Πολιτικής για το 2018-2021. Τέλος, υπάρχουν και άλλα θέματα που συζητήθηκαν στην ΚΟΖΗ και αν μου επιτρέπετε θα αναφέρω πολύ σύντομα δύο θέματα που θα συνεχίσουν να μας αποσχολούν και στην ε, επόμενη Προεδρία. Η διεξοδική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις στατικές προτεραιότητες όπου υπήρξε ερωτηματολόγιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συζητήσαμε στην Κόζη με τα κράτη-μέλη Και ξέρετε ότι ήρθε και ο Επίτροπος Κίνγκ στην άτυπη της Κόζη στη Μάλτα. Και περιμένουμε τώρα την τελική υποβολή έκθεσης που ελπίζουμε ότι θα ε, μας φτάσει την επόμενη εβδομάδα. Σχετικό με αυτό, η κόζη έχει οργανώσει αρχική ανταλλαγή απόψεων για την ε, ε, αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ασφάλεια τον Απρίλιο στα πλαίσια της Προεδρίας της Μάλτας η συνολική, η σφαιρική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα σημαντικό εργαλείο και βάση για τις συζητήσεις μας. Πρόεδρε, μάλλον μακρηγόρησα λίγο. Και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω στην Επιτροπή σας. Uh, Ευχαριστούμε και εμείς. Θα ήθελα να ακούσω τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών με την σειρά που ζήτησαν τον λόγο. Ο κύριος Κουέλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Μήνες μετά την ε, έγκριση της έκθεσής σας, ε, δυστυχώς το θέμα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Ε, και χθε είχαμε ακόμα μια τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλε. Ε, χαίρομαι που το Κοινοβούλιο θέλει περισσότερη και πολεμά για περισσότερη ασφάλεια. Χρησιμοποιούμε καλύτερα το ε, σύστημα ενημέρωση του Σέγγεν, ΣΥΣ, και αυτά τα λέει η έκθεση. Ειδικά σε ό,τι αφορά του ξένου μαχητέ. Είναι απίστευτο που τα κράτη-μέλη δεν δημιούργησαν ένα σύστημα ε, προειδοποίηση και δεν χρησιμοποίησαν το ΣΥΣ για να έχουν περισσότερο και καλύτερο έλεγχο. Και παρότι ότι υπάρχουν αναφορές να αυξηθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ της, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι το κόζι θέλει ε, και προωθεί την καλύτερη χρήση ε, των ισχυών των συστημάτων πληροφοριών παρά τη δημιουργία νέων συστημάτων. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή τροποποιούμε το ΣΥΣ και ε, σύντομα θα έχουμε και τη EuroDAC και ελπίζουμε και το ΕΤΙΑΣ θα είμαστε τότε σε θέση να συζητήσουμε την διαεπιχειρησιακότητα όπως πρέπει και να εντοπίσουμε τα κενά στην στρατηγική για τις πληροφορίες. Ποιες είναι οι απόψεις του Κόζη για αυτό το θέμα. Ε, έχετε κάνει κάποια βήματα, αν έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, σε κάποια φάση μιλήσατε και παραθέτω ενισχυμένη εφαρμογή του πλαισίου Σέγγεν. Τέλος της παράθεσης. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη μελέτη για την ασφάλεια και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ασφάλειας αυτής. Κυρία Σίπολτ. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα της αύξησης, ελπίζουμε, της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Το Κοινοβούλιο πολύ συχνά παραπονιέται για την έλλειψη συνεργασίας και την ε, επαρκή ανταλλαγή πληροφοριών. Αν κοιτάξουμε στο ιστορικό του θέματος, θυμάμαι όταν ε, για πρώτη φορά το 2009 στο Κοινοβούλιο ξεκινήσαμε ήδη να εναρμονίσουμε το ποινικό δίκαιο. Παράλληλα όμως είχα την εντύπωση ότι το ενδιαφέρον το είχαν τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση του εγκλήματος και σπάνια ζητούσαν συνεργασία. Άλλαξε το πράγμα πέρυσι, ειδικά λόγω τρομοκρατίας. Γιατί παρότι πολλά κράτη-μέλη έχουν εμπειρία από τρομοκρατικές επιθέσεις, ε, αυτή η μορφή τρομοκρατίας είναι η πρώτη φορά όπου οι πηγές δεν είναι δεν βρίσκονται σε το εθνικό επίπεδο, αλλά σε εξωτερικό επίπεδο και υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί λόγοι για να συνεργαστεί κανείς. Και βεβαίως πρέπει, μια και θέλουν να συνεργαστούν διάφοροι φορείς και υπηρεσίες, χρειάζεται χρόνος για να υπάρξει αυτή η αλλαγή της νοοτροπίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ ε, θετική η πληροφόρηση που μας δώσατε όταν στην αρχή της παρέμβασής σας μιλήσατε για την αυξημένη χρήση του ΣΥΣ και, την, και τον αυξημένο αριθμό προειδοποίησεων, alert, που εκδόθηκαν. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη δίνουν ε, στο ΣΥΣ, τροφοδοτούν το σύστημα ΣΥΣ, μόνο με τα απαραίτητα στοιχεία. Πιστεύω λοιπόν ότι το ΣΥΣ είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Ε, η γνώση που έχουμε αυξάνει, αλλά και η ετοιμότητα για την ανταλλαγή προφοριών επίσης αυξάνεται. Επίσης, να επανέλθω στο εξή. Η κατάσταση στα κράτη-μέλη και σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα, ε, το διασυνοριακό έγκλημα και το διασυνοριακό έγκλημα, ε, διαφέρει πάρα πολύ. Επομένως, δεν μπορούμε να περιμένουμε το ίδιο επίπεδο πληροφοριών από όλα τα κράτη-μέλη. Να κάνω δύο ερωτήσεις σε εσάς τώρα. Συμφωνείτε ότι υπάρχει μια αλλαγή στη συμπεριφορά των κρατών μελών και των διαφόρων φορέων και οργανώσεων για να χρησιμοποιούν καλύτερα τις πληροφορίες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες καλύτερα και να συνεργάζονται πιο πολύ. Δεύτερη ερώτηση. Θεωρείτε ότι σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα και το διασυνοριακό έγκλημα, ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερες κοινέ ε, ομάδες ερευνητικές ή είναι μια χαρά η σημερινή κατάσταση. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις μετά από τις πολλαπλές επιθέσεις που είχαμε, τρομοκρατικές επιθέσεις. Υπάρχουν παράπονα από το κοινό, αλλά και από πολιτικούς. Και το ερώτημα είναι, γιατί έγιναν αυτές οι επιθέσεις, μια και ξέραμε τον θήτη. Κάποια στιγμή όμως οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα πρέπει να παρακολουθήσουν ε, ή όχι ένα άτομο. Ε, συχνά προκύπτει ότι ήταν μικροεγκληματίας αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Ε, το άτομο αυτό ήταν γνωστό, με κάποια στιγμή ριζοσπαστικοποιήθηκε, αλλά δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι το άτομο αυτό σκόπευε να ξεκινήσει τρομοκρατικές επιθέσεις. Μπορείτε λοιπόν να σχολιάσετε λιγάκι το θέμα αυτό. Ε, δηλαδή να πούμε ότι μια και δεν είναι πάντα τόσο εύκολο ε, να καταλάβουμε από κάποιον ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές ε, ότι θα ριζοσπαστικοθεί τι άλλες ε, πληροφορίε και στοιχεία πρέπει να λάβουμε υπόψη μα για να αποφασίσουμε αν θα παρακολουθήσουμε ή όχι το συγκεκριμένο άτομο τελικά. Ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι Πρόεδρε του ΚΟΖΗ. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα για τη διαχείριση των συνόρων και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, το χώρο δηλαδή της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Φυσικά, αυτή είναι μια θαυμάσια δήλωση προθέσεων. Πολύ ωραία. Όμως, για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζονται διάφορα πράγματα που δεν είναι και τόσο εύκολα. Τι χρειάζεται. Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Σοβαρές. Να ξεκινήσουμε το Ιούλης ή Να του δώσουμε νέες αρμοδιότητες και να του δώσουμε μεγαλύτερο προπολογισμό. Χρειάζεται να καθορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα και χρειάζεται φυσικά χρειάζονται χρήματα στον επόμενο προπολογισμό. Δηλαδή, ο ε, όλοι οι προϋπολογισμοί στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να είναι μεγάλοι. Πετε μου την άποψή σα για τι μετα... Ε, νομοθετικές ε, μεταρρυθμίσεις, για τον νέο ρόλο του EU-LISA και για τον προϋπολογισμό. Τώρα, για τις προτεραιότητες του ΣΟΚΤΑ και το, τις υπόλοιπες. Αναφέρατε διάφορες. Κάτι, υπάρχει κάτι που λείπει από τις αναφορές σας. Ε, καταπολέμηση της παραχάραξης του Euro θεωρούνται δηλαδή διάφοροι ότι δεν παραχαράσετε πλέον το, ευρώ. Εγώ νομίζω ότι ναι. Παρακαλώ, θα μπορούσατε να μου απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις που σας υπέβαλα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Κόζη για την παρουσίαση που μας έκανε. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ Μα μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπατε για την ανταλλαγή πληροφοριών, για τη διαλειτουργικότητα, καθώς και το πρόγραμμα προτεραιοτήτων για την επόμενη τετραετία. Ο κύριος Διαδεμέρα εντόπισε μια έλλειψη, ίσως λείπουν και άλλα πράγματα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ε, σωματεμπορία, τη διακίνηση ανθρώπων, ε, την ε, σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων, ε, που γίνεται και μέσω του ίντερνετ, ε, παιδική πορνογραφία στο ίντερνετ, δηλαδή online, όλα αυτά τα εγκλήματα. Νομίζω ότι είναι εγκλήματα που χρήζουν τη μέγιστη προσοχή μα και θα πρέπει να εντάσσονται στι προτεραιότητε, γιατί μιλάμε για τα πιο α, ευάλωτα θύματα, του πιο μικρού, του πιο νέου. Εσεί αναφέρατε, βεβαίω το ξέρουμε από τι προηγούμενε παρεμβάσει που αναφέρθηκαν σε αυτό, είπατε ότι οι δραματικές τρομοκρατικές ε, επιθέσεις που έπληξαν κάποιες από τις χώρες μας έδωσαν μια νέα όθηση στη συνεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Όμως, να σας ρωτήσω το εξής. Σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, περί, ας πούμε περιβαλλοντικά εγκλήματα, εγκλήματα με και επίκαιρο τα ναρκωτικά από τις έρευνες που είδαμε, ε, υπάρχει σχέση με τα τρομοκρατικές επιθέσεις. Παραδείγματο χάρη, οι, τρομοκρα... τρομοκράτες χρησιμοποιούν ψεύτικα έγγραφα που του τα έδωσαν ποιο, οι εγκληματικέ οργανώσει. Αυτό συνέβη, α πούμε, στη δική μου περιοχή, στην Καμπανία. Αυτή η επιτάχυνση, αν θέλετε να την πούμε έτσι, στην ε, ανταλλαγή πληροφοριών δεν αφορά μόνο την τρομοκρατία, αλλά αφορά και τα εγκλήματα, το οργανωμένο έγκλημα. Ναι ή όχι. Και αν όχι, για ποιο λόγο δεν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί μια και όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία αναφέρατε έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, προέρχονται από τέτοιου τύπου οργανώσεις. Ε, πώς μπορούμε Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα εγκλήματα και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και για αυτού του τύπου τα εγκλήματα, δηλαδή το οργανωμένο έγκλημα. Ο Υπουργό να απαντήσει. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ε... Και ελπίζω να μην ξεχάσω τίποτα. Δεν είναι εύκολο. Θα σας απαντήσω με βάση την εμπειρία που έχουμε, την επιχειρησιακή εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, γιατί όλες αυτές οι πρωτοβουλίε προωθούνται ούτω ώστε να βελτιώσουν και να ενισχύσουν το επιχειρησιακό δυναμικό. Μιλάμε λοιπόν για τους ξένους μαχητές, το σύστημα ΣΥΣ. Το ΣΥΣ είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εργαλείο που αποδείχθηκε αποτελεσματικό. Και το αποδεικνύουν και οι ολοένα και περισσότερες στατιστικές κάθε χρόνο. Τα αποτελέσματα του ενημερωτικού συστήματος του Σέγγεν, του ΣΥΣ, είναι τα υψηλότερα, τα πιο σημαντικά ε, τα τελευταία χρόνια αν λάβουμε υπόψη μας την εποχή από την οποία ιδρύθηκε το ΣΥΣ. Επίσης, οι ξένοι μαχητές. Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις πρέπει να εντοπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα δεν είναι να μπουν τα ονόματα απλώς στο ΣΥΣ ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Δεν είναι αρκετό να ξέρουμε τα ονόματα των ανθρώπων αυτών. Θα πρέπει να έχουμε και αποδεικτικά στοιχεία στα συστήματα. Πολλές φορές έχω αναφέρει, ο, και εσείς το είπατε, ότι κάποιοι άνθρωποι διαπράττουν κάποια δικήματα. Και πολλές φορές ήταν γνωστοί οι άνθρωποι αυτοί στις αστυνομικές αρχές. Αυτό δεν είναι την εντύπωση λοιπόν ότι κάτι δεν κάνει καλά η αστυνομία. Ότι δεν έκανε το καταδύναμη ούτως ώστε να παρεμποδίσει αυτά τα εγκλήματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι υπάρχουν και όλα τα δικαιώματα που έχει το άτομο. Είναι αδύνατον ένας ύποπτος ο οποίος ε, έχει διαπράξει τέτοια εγκλήματα να μπει σε ένα σύστημα ή να μπει ε, σε, ένα, πρόγραμμα επιτήρησης επαορίστο. Δεν γίνεται. Πολλά από τα άτομα αυτά εξάλλου που διέπραξαν τέτοιου τύπου τρομοκρατικά εγκλήματα ήταν γνωστά εδώ και καιρό από την αστυνομία για σοβαρά ή λιγότερα σοβαρά εγκλήματα. Και σας διαβεβαιώνω ότι στις ε, διάφορες επιχειρήσεις και έρευνες λαμβάνουμε υπόψη μας και τα δικαιώματα του ατόμου. Δεν είναι δυνατόν να επιτηρούμε ένα άτομο Και ακόμα και αν συλληφθεί το άτομο αυτό, κάποια στιγμή θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος, γιατί υπάρχουν τα δικαιώματα αυτά σε όλες τις χώρες μας. Γι' αυτό ακριβώς οι αστυνομικές αρχές και οι υπόλοιπε διοκτικέ αρχές συνεργάζονται ούτω ώστε όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται να αξιολογούνται και το προφίλ είναι σωστό, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ποια είναι τα άτομα τα οποία πρέπει να ελέγχονται και να είναι υπό παρακολούθηση συνεχώς και ποια όχι. Επίσης, ανέφερα και το αιτίας ή αναφέρατε και εσείς το αιτίας. Είναι μια άλλη βάση δεδομένων Ε, είναι διαλειτουργικό με το σύστημα ε, εισόδου-εξόδου, entry-exit. Είναι συστήματα που υπάρχουν και στους αστυνομικούς και στις ε, αρχές των επιφύλαξης των συνόρων και πιστεύω ότι η μακροπρόθεσμα θα δώσουν και περισσότερα αποτελέσματα από αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό επίσης ότι υπάρχουν και αρκετές χώρες οι οποίες εφαρμόζουν αυτά τα συστήματα. Προσπαθούμε να έχουμε ομοιομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούν και υπάρχουν αυτά τα συστήματα σε όλες τις χώρες, παντού. Εν συνεχεία, τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι προειδοποίησεις του συστήματος ΣΥΣ. τα εργαλεία για τη βελτίωση της ε, ασφάλειας της προστασίας και της προστασίας των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τέτοιες πρωτοβουλίες και όταν το κάνει, αυτό που θέλει είναι για κάθε πρόταση να υπάρχουν πάντα τα εργαλεία, ούτω ώστε και η προστασία των δεδομένων, αλλά και η χρήση και διάδοση των πληροφοριών γίνεται, ούτως ώστε να μην ε, καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλες αυτές οι προτάσεις ε, προωθούνται παράλληλα. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οποιοδήποτε πρέπει να ελεγχθεί με βάση τα στοιχεία που έχουμε στις βάσεις δεδομένων, ελέγχεται. Και αυτό το επιτρέπει η νομοθεσία η οποία πρέπει να είναι επαρκώς αυστηρή, ούτως ώστε να εξασφαλίζει ότι παράλληλα και τα δικαιώμα, δικαιώματα του ατόμου αυτού δεν καταπατώνται. Ε, The same thing is uh, on information exchange. Το ίδιο και για την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών Συχνά η ανταλλαγή πληροφοριών μέχρι τώρα γινόταν σε διμερή βάση. Τώρα όμως πια ε, ανοίγει το πλαίσιο. Εμείς, ε, ο κόσμος είναι πάρα πολύ μικρός και η Ευρώπη είναι ακόμα μικρότερη. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει κάποιο σύστημα είναι διαθέσιμη και στις υπόλοιπες ε, διοκτικές αρχές. Και φυσικά οι διατάξεις για διασφάλιση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών δικαιωμάτων, γίνονται σεβαστές. Βλέπουμε όμως μία αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών, ένα επιμερισμό των πληροφοριών και αυτό θα παραμείνει προτεραιότητα. Γι' αυτό έχουμε αυτό το νέο εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα. Και ελπίζουμε να αυξηθεί αυτή η τάση, ούτως ώστε όλες οι διοκτικές αρχές να έχουν τα εργαλεία που περιμένουν. Από πείρα σας λέω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών ε, για τέτοιου είδους ανθρώπων είναι η βάση για την, ε, τις έρευνες και για την επιτυχή καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Η διαλειτουργικότητα και οι ανταλλαγέ πληροφοριών είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του ΚΟΖΗ αυτή τη στιγμή. Ασχολούμαστε εδώ και καιρό με αυτό το, πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει και ένας οδικός χάρτης, υπάρχουν 50 πρωτοβουλίες που πρέπει να προωθήσουμε. Το πράγμα προχωράει ομαλά. Ελπίζουμε να σημειώσουμε επιτυχία για τους ανθρώπους που υπηρετούμε, αλλά και για να σημειώνουν ακόμα περισσότερες επιτυχίες οι διοκτικές μας αρχές. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε και τις καλύτερες νομικές ε, διατάξεις, ούτως ώστε να εφαρμόζονται σωστά αυτές οι προτάσεις. Σας διαβεβαιώ ότι έτσι θα γίνει. θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και το σωστό προπολογισμό, τον απαραίτητο προπολογισμό για να είναι λειτουργικό το σύστημα. Έχουμε ετοιμάσει ήδη αυτόν τον οδικό χάρτη. Θέλουμε να έχουμε και το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα, ούτω ώστε το σύστημα να εφαρμοστεί. Ε, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και με την eu ε, που είναι ο πρωταγωνιστής στα παρασκήνια πίσω από αυτό το σύστημα. Κάποιος ευρωβουλευτής ανέφερε την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Ναι. Είναι μία από τις δράσεις στα πλαίσια του policy cycle, του κύκλου πολιτικής και της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος. Δεν το ξεχάσαμε, ήταν και στο παρελθόν προτεραιότητα και θα εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει προτεραιότητα. Δυστυχώς το πρόβλημα αυτό είναι όλο και πιο σημαντικό. Δεν μιλάμε μόνο για διακίνηση και σωματεμπορία ανθρώπων, αλλά κυρίως παιδιών και θα πρέπει να τύχει της δέουσας προσοχής. Όταν μιλάμε για τις προτεραιότητες δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε εδώ, δεν υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, αλλά αυτές είναι οι κύριες προτεραιότητες μετά από τις, που καθορίστηκαν μετά από τις αξιολογήσεις που έγιναν μετά από τον πρώτο κύκλο πολιτικής. Θελήσαμε να βελτιώσουμε τις ε, προτεραιότητες των ετών 2018-2021 ούτως ώστε να παραμείνει προτεραιότητα η καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Επίσης, η παραχάραξη και τα ψεύτικα έγγραφα. Ε, η παραχάραξη του ευρώ είναι κάτι που εξακολουθεί να υπάρχει. Το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε ως πρώτη προτεραιότητα σε αυτή την έκθεση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να συλλέγουμε πληροφορίες και να διαθέτουμε εργαλεία για να καταπολεμούμε και τέτοιου τύπου αδικήματα. Επομένως, ε, δεν υπάρχουν μόνο οι προτεραιότητες για την καταπολέμηση του εγκλήματος που ανέφερα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με όλες τις ε, διοκτικές αρχές, ακόμα και σε διμερή βάση μερικές φορές, ούτως ώστε όλες οι διοκτικές αρχές, κάθε διοκτική αρχή να έχει ε, τα απαραίτητα εργαλεία στην, ε, στα χέρια της για να, καταπολεμεί όλα, να καταπολεμάει όλα τα είδη του εγκλήματος και την τρομοκρατία. Ξέρετε ότι διανύουμε πολύ ζωφερές εποχές, γιατί το είδος των τρομοκρατικών επιθέσεων που λαμβάνουν χώρα τώρα είναι επιθέσεις που δεν τις είχαμε φανταστεί στο παρελθόν. Δεν φανταζόμασταν ότι τα οχήματα θα χρησιμοποιούνται τόσο ε, συχνά ως ε, όπλα. Το ίδιο. Το ίδιο λοιπόν ε, ισχύει και για του αλλοδαπού μαχητέ. Όχι μόνο για του τρομοκράτε μαχητέ, αλλά ξέρουμε ότι το πρόβλημα αυτό θα συνεχίσει να διαγκώνεται. σε ό,τι αφορά τους ροδαπούς τρομοκρατές μαχητές. Ξέρουμε και τι συνέπειες θα έχει αυτό. Και για τις οικογένειές τους. Μιλάμε για νεαρά άτομα τα οποία δεν έχουν γνωρίσει τίποτα άλλο παρά τον πόλεμο, δεν ξέρουν κάτι άλλο. Και λαμβάνονται και προβαίνουν σε επιθέσεις κατά των κρατών τους. Ελπίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σέλλα. Και έτσι με την παρεμβάση της ε, ΚΟΖΗ ολοκληρώνονται κάποια ζητήματα όπως το θέμα της λειτουργικότητας, της ανταλλαγής πληροφοριών. Προφανώς είναι θέμα το οποίο θα συνεχίσει να παραμένει στην ατζέντα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση της ΚΟζη, πολύ ευπρόσδεκτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας ε, εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους που ήταν πολύ εντελεχείς και να περάσουμε στο επόμενο θέμα το οποίο είναι η παρουσίαση της Προεδρίας του Συμβουλίου για την ιστορικό ελέγχο, τον έλεγχο συγγνώμη, των ιστορικών συνόρων. 11 Μαΐου, στις 11 Μαΐου του 2017 το Συμβούλιο έκρινε μια περαιτέρω εφαρμοστική απόφαση με σύσταση να παραταθούν οι προσωρινοί ιστορικοί έλεγχοι που επιτρέπουν στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Σουηδία και την Δανία να παρατείνουν για μέγιστη περίοδο 6 μηνών τους εσωτερικούς ελέγχους. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην Μαλτέζικη Προεδρία για την παρουσίαση της εφαρμοστικής απόφασης και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει τις απόφασεις για πρόταση με τι συστάσει του Συμβουλίου και μετά θα γίνει συζήτηση. Θα ξεκινήσει η συζήτηση. Η Μαλτέζικη Προεδρία λοιπόν πρώτα. Δεν ξέρω, ήταν η κυρία Κάκ, η Άλσον Κάκ ή κάποιος άλλος. Αν θα θέλετε παρακαλώ να, σας, να μας πείτε ποιο θα κάνει την παρουσίαση. Όχι, ο συναδελφό μου ήταν να, να την κάνει. Όπως ξέρετε, τον Μάιο 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια σύστοση για την τρίτη και την ε, τελευταία παράταση εξαμήνου. Η πρόταση αυτή συζητήθηκε με το Συμβούλιο σε τεχνικό επίπεδο και στο Κορυπέρ. Το Συμβούλιο επιτέλεσε σημαντική πρόοδο και ε, μάλλον επένεσε για την προ... σημαντική πρόοδο που έχει επιτελεστεί ε, από τις προηγούμενες συστάσεις και σε πολλά μέτωπα. Βεβαίω, πέραν αυτού, το Συμβούλιο συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η κατάσταση δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα και ότι η σύσταση για την παράταση των ελέγχων πρέπει να εγκριθεί. Η εκτελεστική απόφαση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 27 Μαΐου 2017, συστήνοντας την παράταση του συστήματος ε, εσωτερικού ελέγχου των συνόρων για έξι μήνες. Έφεραν αντιρρήσεις κάποια κάτι μέλη, αλλά όπως τα είδατε η εκτελεστική απόφαση ακολουθεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολύ στενά. Επίσης υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι όπου δει, όπως προβλέπει η νομοθεσία, προκειμένου να αποφευχθούν οι εσωτερικοί έλεγχοι στα σύνορα. Αυτό θα πρέπει να είναι η λύση εσχάτου καταφυγίου. Μετά από διαβουλεύσεις και συνομιλίες με όμορα κράτη-μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο συζήτησε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επιτόπιους ελέγχους, κάτι που ε, έγινε επίσης ευπρόσδεκτο. Okay, and, um, and now the Commission. Ευχαριστούμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέκαθεν ήταν να υπάρχει μια ε, ε, εύρυθμο λειτουργούσα περιοχή Σέγγεν, χώρο Σέγγεν, ε, χωρίς εσωτερικούς ελέγχους. Να πω τώρα τι γίνεται με τους εσωτερικού ελέγχους στα σύνορα και τι γίνεται και με τη σταδιακή κατάργησή τους. Ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την παράταση για ένα τελευταίο εξάμεινο ήταν η παρουσία μεταναστών στην Ελλάδα και οι πολύ αργές μετακινήσεις μεταναστών στη λεγόμενη οδό Βαλκανίων. Επειδή όμω χρειάζονται περισσότερε προσπάθειε όπω εντόπισαν και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και όπω εντοπίστηκε στην 13η ε, έκθεση της 18ης Ιουνίου ή μετεγκαταστάσεις και επιστροφές από την Ελλάδα θα πρέπει να ε, εντατικοποιηθούν και να ισχύσουν πλήρως πάλι όλοι οι κανόνες. Επειδή αυτή θα είναι η τελευταία παράταση, να πούμε ότι η έλεγχη στα σύνορα θα πρέπει να είναι ε, έκτακτη μόνο ε, και κατεξαίρεση και ως μέτρο τελευταίου σκάτου καταφυγίου. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, και εδώ θα ήθελα να δοθεί έμφαση, τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέτρα με παρόμοιο ε, αποτέλεσμα όπως η εσωτερική έλεγχη. Η Μαλτέζικη Πρεδρία ήδη ανέφερε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει οι αστυνομικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν ε, περαιτέρω τις τους πόρους τους για να είμαστε αποτελεσματικοί και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς τους ελέγχους παρά στους έλεγχους στα εσωτερικά σύνορα. Κατά την άποψή μας δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν και αστυνομικοί έλεγχοι και ε, έλεγχοι σύνορου στα σύνορα, αλλά η ουσία είναι να αντικατασταθούν οι έλεγχοι στα σύνορα από τους αστυνομικούς. Εφόσον όλα αυτά λειτουργήσουν, θα έχουν πολύ περισσότερο νόημα και λογική, γιατί θα υπάρχει περισσότερη ευελιξία για τις αρχές ελέγχου θα μπορούν να κάνουν τους ελέγχους τους δρόμους ε, μετακίνησης και διέλευσης λόγω χάρη, μετακόμισης, όχι μόνο να κάθονται στα σύνορα και να περιμένουν εκεί. Κάτι που στην, τελική, στην, στην ουσία είναι σπατάλη πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει την σύσταση για τους αστυνομικούς ελέγχους όσο το δυνατόν συντομότερα και το αργότερο μέσα στο εξάμεινο αυτό, ε, την τελευταία παράταση δηλαδή στο Νοέμβριο, οργανώνουμε τώρα ένα εργαστήριο με τη συμμετοχή των 10 πλέον ε, ε, ε, ε, άμεσα μάλλον εμπλεκόμενων κρατών μελών ε, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου με σκοπό να υπάρξει μια επιτάχυνση της αστυνομικής συνεργασίας ήδη από το Σεπτέμβριο. Θέλουμε να συζητήσουμε ήδη με τα κράτη-μέλη πώς θα οργανωθούμε. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ανέφερα την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε πλήρω στην κανονική κατάσταση του Σέγγεν στο τέλο τη χρονιά. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ που για την δική σα συνεισφορά. Εγώ να επιστολή προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο, ζητώντα εκθέσει ε, αναχώρα, στοιχεία αναχώρα. Δεν έλαβα καμιά απάντηση. Ευχαριστώ. Ναι, να σας δώσω μια απάντηση καταφατική ε, Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει πλήρω το τιμά σα, όμω η Επιτροπή δεν είναι εκείνη που συντάσσει τι σχετικέ εκθέσει. Ήρθαμε σε επαφή με όλα τα κράτη-μέλη του Σέγγεν ε, που αφορούσε το ερώτημά σα, του ρωτήσαμε και αν συμφωνούν να ε, μοιραστούν οι εκθέσεις αυτές και στο Κοινοβούλιο και περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Μόλις έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων ε, κρατών μελών, αμέσως θα σας στείλουμε τις σχετικές εκθέσεις, όλες τις εκθέσεις, σε εσά το Ευρωκοινοβούλιο. Αμέσως τι εννοείται. Σας έγραψε το Μάιο αφού σας λέω, περιμένουμε να απαντήσουν τα κράτη-μέλη. Δεν είμαστε εμεί αυτοί που συντάσσουμε. Ναι, το ξέρω, ε, το ξέρω, αλλά ε, χρειάζεται η συμφωνία των κρατών μελών. Το συζητήσαμε και με τι νομικέ μας υπηρεσίε. Μα δεν σας λέω, όχι, περιμένουμε, το ok από τα ενδιαφέρομενα κατήμελη. Ναι. Μόλι μα απαντήσουν, θα σα το στείλουμε. Ναι, κοιτάξτε, πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο που το γυρνάτε σε μένα το μπαλάκι, αλλά ξέρετε, ξέρω πολύ καλά δεν είστε συντάκτε των εκθέσεων αυτών. Εγώ θα ήθελα τουλάχιστον να είχατε την ευγένεια να μου γράψετε και να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει mm. Και είναι σημαντικό να είναι ενήμεροι και ευρωβουλευτέ για το τι ακριβώ συμβαίνει εντωμεταξύ. Αμέσω, ε, από το Μάιο δεν είναι αμέσω. Τι θα πει αμέσω. Σήμερα ή σε πέντε χρόνια. Χρησιμοποιήστε μια πιο φυσιολογική γλώσσα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Να ακούνε και ευρωβουλευτέ. Αμέσω σημαίνει ότι θα τα δούμε κάποια στιγμή αυτά τα στοιχεία. Ιδάλω θα ζητήσω από τον Επίτροπο να μου στείλει ένα κείμενο αμέσω. Αυτό θα πει αμέσω. Η κυρία Γκραπίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτά που είπε το Συμβούλιο, παρά το γεγονό ότι μιλάμε με κάποιον διαφορετικό πλέον. Δεν είναι το ίδιο άτομο που μας παρουσίασε τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι μία από τις προτεραιότητες ήταν να βελτιωθεί η βάση του ΣΕΝΙΕΝ και ο τρόπος λειτουργίας της. Εγώ συμμετείχα σε όλες τις συζητήσεις για θέματα εσωτερικής ασφάλειας στα πλαίσια του Σένιεν. Και στη χώρα μου διαρκώς ο κόσμος με ρωτάει γιατί η χώρα μας, η Ρουμανία, δεν είναι μέρος της ε, του Σέγγεν, ενώ η χώρα μας πληρεί όλες τις ε, προδιαγραφές. ή ταξιδιώτες, όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ασφάλεια της, θα πρέπει να μιλάμε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πρόκειται για χώρες Σέγγεν είτε όχι. Και εγώ νομίζω ότι στην ε, Ρουμανία η κατάσταση ό,τι αφορά την ασφάλεια είναι πολύ καλύτερη από ό,τι σε κάποιες χώρες του Σέγγεν. Δεν έχουμε προβλήματα τρομοκρατίας, Και έχουμε και το ίδιο πρόβλημα με εσά, με τη Μάλτα, όπω και με τι προηγούμενε προεδρίε. Δεν λαμβάνουμε απαντήσει. Δεν μα απαντάει ούτε το Συμβούλιο ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δεν υπάρχει ένα ενίο εξωτερικό σύνορο ω περίμετρο ασφαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ τι θα το και πάλι αυτή την ερώτηση, ελπίζοντα μήπω πάρω μια απόφαση σήμερα τουλάχιστον. Νομίζω ότι αν η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Σουηδία πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους ε, συνοριακούς ελέγχους, ε, τότε ναι, μπορούν να υπάρξουν επιπρόσθετα μέτρα. Αλλά τι γίνεται μετά από έξι μήνες. Ε? Θα συνεχίσουμε να παρατηρούμε διαρκώς κατά έξι μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Έλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το έχω πει και ξανά και ξανά. Και έχω πλέον την αίσθηση ότι το Συμβούλιο μαζί με την Επιτροπή όντως κάτι μας κρύβουν. Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε τους ιστορικούς ελέγχους. Έχουν περάσει ένα έτος α, από τότε που και κάποιες χώρες αποφάσισαν να εισαγάγουν ιστορικούς ελέγχους και περίπου έξι μήνες από τότε που παρε, πέρασε η προθεσμία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμφωνία του Συμβουλίου να σταματήσουν αυτοί οι έλεγχοι. Και είναι ανησυχητικό ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει στη διάθεσή του όλε τι πληροφορίε που χρειάζονται. Δεν υπάρχουν σχετικέ πληροφορίε, Δεν μα έχουν αποσταλεί όλε οι απαραίτητε πληροφορίε. Και θα θυμάστε ότι έχω θέσει το ερώτημα στην Επιτροπή μα. Πώ μπορούμε να αξιολογήσουμε αν χρειάζονται όντω έλεγχοι, αν δεν έχουμε πληροφορίε στη διάθεσή μα. πόσους ε, παράνομους μετανάστες σταματήσαμε, τι είδη ελέγχων έχει γίνει, ποιος είναι ο οικονομικός αντίκτυπος των ελέγχων και τον περασμένο μήνα σε επίστολη προς τον Επίτροπο και προς ε, τον πρόεδρο της Επιτροπής αναφέραμε αυτά που είπατε πριν από κάποια λεπτά. Τώρα ζητώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιαστεί στην Επιτροπή για τα, το Σένιεν για να μας παρουσιάσει τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο πολύ διαφάνεια το θέμα αυτό. Τέλος, Πρόεδρε. Ακούσαμε ότι είτε η Μαλτέζικη Προεδρία, είτε μάλλον και η Μαλτέζικη Προεδρία και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλούν για αστυνομικούς ελέγχους. Δεν έχω πρόβλημα με τους αστυνομικούς ελέγχους και πιστεύω ότι πραγματικά χρειάζονται πιο έξυπνοι, αν θέλετε, και στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι. Αλλά είδα ένα έγγραφο το οποίο διέρευσε, έγγραφο της Προεδρίας, όπου παραθέτω γίνεται λόγος για εντατικοποίηση αστυνομικών ελέγχων σε όλη την ε, επικράτεια. Είναι πρόσφατο το έγγραφο, μια εβδομάδα. Το ερώτημα λοιπόν που έχω είναι το εξή. Το Συμβούλιο τι προετοιμάζει από αυτή την άποψη, τι έχετε ακριβώς υπόψη όταν μιλάτε για εντατικοποίηση αστυνομικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια. Η Επιτροπή αυτή χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια για το Σέγγεν. Το Σέγγεν είναι πολύ α, ε, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες, τους οποίους και εκπροσωπούμε σας, θυμίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πρόεδρος. Ξέρετε ότι Προεδρία έχει εμπειρία στο θέμα αυτό. Θα ζητούσα από την Προεδρία να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καλέσει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις. Η κυρία Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες που μου δώσατε. Το 2015 στην Σουηδία γίναμε μάρτυρες μιας μαζικής ε, μετανάστευσης και υπήρχαν έλεγχοι στα σύνορα. Χρειάστηκε όμως αρκετός χρόνος για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτούς τους έλεγχους στα σύνορα. Αν δεν είχαν γίνει αυτοί οι έλεγχοι εξαιτία αυτών των μεταναστευτικών ροών θα είχε καταρρεύσει η χώρα μου. Τώρα έχουμε ελέγχου στα σύνορα και εγώ είμαι πραγματικά ευγνώμων γι' αυτό. Αλλά όπως υπόθηκε αυτή είναι η τελευταία παράταση των ελέγχων στα σύνορα. Εν τί αυτή περιπτώσει ε, είναι σαφές ότι ένας από τους πυλώνες της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη θα αποκατασταθεί το Νοέμβριο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μια σειρά από μετανάστες που φτάνουν, φρέσκοι μετανάστες που φτάνουν στην Ιταλία. Και ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν πρόκειται να μεταρρυθμιστεί φέτος, παρά τις ε, μαζικές αυξήσεις των ε, μεταναστών. Διερωτώμε λοιπόν πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια περαιτέρω μεταναστευτική ροή τη στιγμή που δεν θα έχουμε πια ελέγχου στα σύνορα. Πώς θα γίνει αυτό. ξεχνάμε ότι χρειάζεται χρόνος για να επιτρέψουμε ελέγχους ε, ή για να γίνουν οι αστυνομικοί έλεγχοι για τους οποίους μιλάμε σήμερα. Εξού και το ερώτημά μου. Ακούσαμε την Κομισιόν να μας λέει ότι θα γίνονται αστυνομικοί έλεγχοι που θα αντικαθιστούν ή θα υποκαθιστούν τους ε, συνοριακούς ελέγχους. Όμως η έλεγχη το 2013 δεν μπορούσαμε να κάνουμε ε, ελέγχους σε μετανάστες στην ε, Σουηδία, γιατί είχαμε μία σειρά από άτομα τα οποία κυκλοφορούσαν στη Σουηδία χωρίς ε, έγγραφα. Πώς θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι για αυτή την περιπτώση. Σας ευχαριστώ κυρία Σατζοντίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι η προηγούμενη φορά με την παράταση Νομίζαμε ότι ήταν πραγματικά η τελευταία παράταση. Τώρα όμω φαίνεται ότι είναι πραγματικά η τελευταία φορά. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι πόσο βέβαιοι είμαστε ότι είναι πραγματικά η τελευταία φορά αυτή. Είναι πολύ πολιτικό το ζήτημα για την λειτουργία του Σέγγεν, των εσωτερικών ελέγχων. Είμασταν περήφανοι. περήφανοι που δεν υπήρχαν αυτή η εσωτερική έλεγχη και φαίνεται ότι πλέον είναι φυσιολογικό να παρατείνονται αυτή η έλεγχη. Η επιχειρηματολογία δεν μου προκαλεί έκπληξη. Μιλάμε για την κατάσταση στην Ελλάδα, τους ε, πρόσφυγες που καταφθάνουν στην Ελλάδα. Η οδός των Βαλκανίων έκλεισε το Φεβρουάριο του 2016. Το Μάρτιο του 2016 είχαμε τη συμφωνία με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το σουηδικό, δανικό σύνορο ή το αυστριακό, γερμανικό σύνορο αντιμετωπίζει προβλήματα με τεράστιες εισρωές και αφήξεις προσφύγων και λαθρομεταναστών. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Θα υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που θέλουν να συνεχίσουν να παρατείνουν τους έλεγχους στα κράτη-μέλη αυτά. Και αν ένας από τους λόγους είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η με την κατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα ή από την Ιταλία, φαίνεται ότι είναι μια κατάσταση διπλού ωφέλου για τα κράτη. Αυτά που δεν θέλουν ούτε με την κατάσταση, ούτε να σταματήσουν οι έλεγχοι για του αστυνομικού ελέγχου. Αυτό το καταπολεμώ στι κάτω χώρε, στη χώρα μου, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν γίνεται δηλαδή έλεγχο στα σύνορα, άρα γίνεται αστυνομικό έλεγχος με δειγματοληπτικούς ελέγχους κάποια χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η δειγματοληπτική έλεγχη γίνεται πάντα σε πινακίδες αυτοκινήτων από την Ανατολική Ευρώπη. Αν αρχίζουμε να κάνουμε σταθερά τέτοιου αστυνομικού ελέγχου αντί για ελέγχου στα σύνορα, τα πράγματα θα δυσκολέψουν παραπάνω. Και είδα παραδείγματα όπου οι Ολλανδική αστυνομία καταδοκούσε σε βελγικά πάρκινγκ για να δουν ποιο θα περνούσε τα σύνορα και μετά με εγώ και να ειδοποιήσει του συναδέλφου από την άλλη πλευρά των σύνορων ότι ο τάδε οδηγό με τι τάδε πινακίδε ε, θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό δεν μετρούσε ω ε, έλεγχο σύνορων, αλλά ω ε, αστυνομικό έλεγχο. Α μην κινηθούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Αν θέλουμε ε, Εσωτερικού ελέγχου α στηρίσουμε τουλάχιστον του κανόνε που υπάρχουν, δηλαδή δειγματοληπτική έλεγχη κάποιε ώρε τη ημέρα. Σχεδόν ολοκλήρωσα λοιπόν την παρέμβαση μου, Πρόεδρε, αλλά πραγματικά για κάτι το οποίο είναι τόσο πολύτιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αντίδραση του Συμβουλίου πραγματικά είναι περιορισμένη και ισχνή. Δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουν τι οικονομικά συμφέροντα παίζονται εδώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω ένα τεράστιο ερωτηματικό ως προς το κείμενο αυτό. Δεν φαντάζομαι, κύριε Κουαλιό, να ε, σας φαίνεται περίεργο. Στη χώρα του αναφέρονται ε, η έλεγχη στα σύνορα ε, αναφέρεται πρώτη δική μου, γιατί εμεί ήμασταν αυτοί που ζητήσαμε την αποκατάσταση του ελέγχου στα σύνορα. Αυτό έγινε τη στιγμή που στην COP21 ε, είχαν συμπέσει και οι επιθέσεις του Παρισιού και συστηματικώς τους ζητούσαμε του τους ελέγχους αυτούς όχι για την καταπολέμηση των μεταναστευτικών ροών αλλά για τις θερμοκρατικές επιθέσεις, την καταπολέμηση της θερμοκρατίας να πω ότι η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει τρομοκρατικέ απειλέ, αλλά νομίζω ότι είναι η μόνη που ζήτησε την αποκατάσταση των ε, εσωτερικών ελέγχων, των ελέγχων στα σύνορα για σκοπούς καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Δεν βλέπω να υπάρχει καμιά συνέπεια, αλλά στην πραγματικότητα η Γαλλία χρησιμοποιεί την αποκατάσταση των σύνορων και για την καταπολέμηση τη λαθρομετανάστευση. και θα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ. διότι αφορά ε, την εκλογική περιφέρεια που εκλέγουμε τον νότο της Γαλλίας, τα σύνορα Γαλλίας-Ιταλίας. Υπάρχουν συστηματικός έλεγχοι και συστηματικός έλεγχοι, όχι για όλους, συστηματική έλεγχη στα σύνορα. Και όχι όπως είπε η κυρία Σαρχεντίνη, όχι μόνο για τα ε, χρώματα, ε, για τις πινακίδες των αυτοκινήτων, αλλά και για το χρώμα του δέρματος. Ε, δηλαδή, εάν τίποτα Γάλλοι έχουν κανένα δέρμα λίγο πιο σκούρο, ή είναι μαυροτσούκαλοι, τους ελέγχουν κατευθείαν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα ε, και άλλα προβλήματα. Όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται οι έλεγχοι σε αυτό το πλαίσιο. Ε, οι πόροι και οι διάφοροι φρουροί που έχουν κατ' εξαίρεση αναλάβει καθήκοντα στην Γαλλία εκτάκτως αυτοί που βρίσκονται στα σύνορα λοιπόν Γαλλίας-Ιταλίας αυτοί κάνουν έλεγχο με σκοπό να καταπολεμήσουν την μετανάστευση εδώ θα πρέπει λοιπόν να αναφέρω ότι όντω μα ανησυχεί η αποκατάσταση των εσωτερικών ελέγχων στα σύνορα Γαλλία-Ιταλία και κύριε Κοελιό, θα σα έλεγα ευχαρίστω να πάμε να κάνουμε μια πολύ μικρούλα αποστολή εκεί στα σύνορα Γαλλία-Ιταλία για να δείτε ότι υπάρχουν κάμποσα προβλήματα. Και όπω ανέφερε και το Συμβούλιο των Υπουργών, θα εγκριθεί ένα νέο πρόγραμμα μέτρων και δράσης κατά της τρομοκρατίας που θα συστηματικοποιήσει την ε, κήρυξη ε, έκτακτης ανάγκης και θα γίνει μια κατάσταση πάγια. Εκεί θα έχουμε νομίζω πολλά να πούμε για τη διασύνδεση μετανάστευσης, τρομοκρατίας και σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών. Πολύ φοβούμαι ότι η χώρα μου που θέλει να θεωρεί τον εαυτό της πατρίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει βιαστεί να υπογράψει τη σχετική χάρτα, θα γίνει και πρωτοπόρος στην ε, οπισθοχώρηση στον τομέα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βεζιά, ο κύριος Ράντοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε η ασφάλεια στο χώρο Σέγγεν και το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εξαρτώνται πολύ από τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα εξωτερικά σύνορα και εξαρτάται από το πώς χώρες όπως η Βουλγαρία με εξωτερικά σύνορα τηρούν πολύ ψηλά πρότυπα για την προστασία των σύνορων ή όχι. Πάντως, αυτό εξαρτάται και από τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους. Εδώ λοιπόν ε, για το χώρο Σέγγεν ε, ένα τεχνικό ερώτημα. Θα γίνει κάτι από το Συμβούλιο για να έχει και η Βουλγαρία πρόσβαση στο σύστημα VIS, το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, αλλά και για το ΣΥΣ ε, βάσει του άρθρου 24. Ευχαριστώ. Κανένα άλλο, λέει ο Να ακούσουμε τι ε, τη της ε, και τη Επιτροπή. παρακαλώ. Θα διαβάσουμε τα μηνύματα και θα βοηθήσουμε και την Επιτροπή να συλλέξει ό,τι στοιχεία χρειάζεται. Προετοιμάζουν τα κρατημέλη διάφορες εκθέσει και θα δούμε τι μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σα. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στην πρακτική ε, συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχω συνδεθεί με τον ε, βοηθό του κυρίου Κόελιο σε διάφορε περιπτώσει και θα ε, αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε μαζί του και θα δώσουμε πληροφορίες. Okay. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ο Πρόεδρος. Να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κάνει αξιολόγηση για το Σέγγεν πριν από κάποια χρόνια, νομίζω το 2012 ήταν, και ε, συμπεράνομαι ότι φυσικά αυτέ οι δύο χώρε είναι έτοιμε για το Σέγγεν. Όπω ξέρετε, ότι είναι είναι μονομερής, είναι ομόφωνη η απόφαση του Συμβουλίου. Όλα τα κρατημέλη πρέπει να συμφωνήσουν και αυτό είναι το θέμα εδώ. Ίσως δεν ήμουν σαφής ε, προηγουμένως. Όταν θα συμφωνήσουν όλα τα κράτη Σέγγεν που είναι σχετικά, τη στιγμή μάλλον που θα υπάρξει αυτή η συμφωνία, θα μοιραστούμε όλες τις ε, μηνιαίες εκθέσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με χαρά. Όπως είπε και ο κ. Κοέλιο, ενδεχομένως όντω, να ήταν σημαντικό να υπάρχει μια συνάντηση και κλεισμένων των θυρών για τα θέματα αυτά. Για να δοθούν και πληροφορίες για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τους αστυνομικού ελέγχου. Να τονίσω ότι από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιδείξαμε τη μέγιστη ευελιξία και προ το Συμβούλιο και προ τα κρατη για το θέμα αυτό. και τώρα είμαστε σε ένα πάρα πολύ περίεργο σημείο σε ό,τι αφορά το άρθρο 29 για την παράταση, γιατί ο κώδικα διεντολογία ε, ορίζει με σαφήνεια ότι έχουμε εξαντλήσει όλες τις ενδεχόμενε παρατάσεις. Μέχρι τον Νοέμβριο λοιπόν δίνεται παράταση, Το Νοέμβριο Ελπίζουμε να έχουν καταλαγιάσει και τα έντονα να έχουν περάσει εκλογέ, να έχει καταλαγιάσει και το κύμα των μεταναστών. Πρόκειται για ένα σημείο καμπή, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την εκ νέου χρήση του Σέγγεν. Κάποιε φωνέ από κράτη-μέλη το κατά πόσον αυτή θα πρέπει να είναι τελική παράταση και αυτό είναι ανησυχητικό προφανώς γιατί μιλάμε για το νομικό πλαίσιο το οποίο πλέον έχει εξαντληθεί 100% και το έχει επαναλάβει αυτό πολλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη ότι οι γενικοί κανόνες για την εισαγωγή εσωτερικών ελέγχων εξακολουθούν να ισχύουν 100% και πάντα ισχύουν. Δηλαδή, ναι, για την Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι εδώ και καιρό τόσο οξύ όσο ήταν. Υπάρχει ένα θέμα για την Ιταλία. Πάντα λοιπόν υπάρχει η, η δυνατότητα να επανεισαχθούν εσωτερικοί έλεγχοι σε άλλα τμήματα των συνόρων για άλλους λόγους. Για δύο μήνες το όριο σε περίπτωση που χρειάζεται άμεση δράση ή για έξι μήνες σε περίπτωση προβλεπόμενων γεγονότων. Τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν πολύ ευελιξία και η Επιτροπή επέδειξε ότι μπορεί να επιδείξει ευελιξία. Δεν μπορούμε όμω να ακολουθούμε διαρκώς την εξαίρεση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επανέλθουμε και στον κανόνα, όπως επεσήμεναν και διάφοροι ευρωβουλευτές. Ε, η εσωτερική έλεγχη είναι πολύ επιζήμια και για τον πολίτη και για την οικονομία και για το Σέγγεν και την επιβίωση του Σέγγεν. Γι' αυτό λοιπόν ε, επαναλαμβάνω και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιδείξει μεγάλη ευελιξία. Με 10 κρατημέλη θα γίνει στις 10 Ιουλίου μια συνάντηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποστείλει ένα ισχυρά αυτό το μήνυμα για το ότι νομικός πώς και λειτουργικός πώς αυτό θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές για τα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ε, θα φτάσουν στα κρατη και ελπίζουμε μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου μπορούμε τον Νοέμβριο να επανέλθουμε στο Σέγγεν. Ελπίζω με τον τρόπο αυτό να κάλεψα τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, δεδομένης της σημασίας του θέματος αυτού, κύριε Κοέλιο, μήπως θα θέλετε να απαντήσετε σε αυτά που ακούσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Προεδρία. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώνω την προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραστεί στην ομαδεργασία σε για το ΣΕΝΙΑ. Την ευχαριστώ. Αλλά να επανέλθουμε στο ζήτημα που μας απασχολεί. Χειροκροτούμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργηθεί ένα οδικός χάρτης για την επιστροφή στο Σέγγεν. Και αυτά που διαπιστώνουμε στην παρούσα φάση είναι ότι κάτι κράτη-μέλη θέλουν να κάνουν παρατάσεις πέρα από το σύνομο με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτό αποτελεί πρόβλημα. Έχουμε κι άλλο ένα πρόβλημα και γι' αυτό αναφερθήκα στα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει από το Συμβούλιο. Από ό,τι φαίνεται, κάποιο στο Συμβούλιο διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα να παραδοθεί περαιτέρω η εισαγωγή, η επανεισαγωγή των εσωτερικών ελέγχων. Και μου φαίνεται ότι προετοιμάζουν έναν τρόπο για να καταπατήσουν το νομικό αυτό πλαίσιο, δημιουργώντας αυτή την εντατικοποίηση των αστυνομικών ελέγχων. Αυτό θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε το ευρωπαϊκό δίκαιο ως έναν τρόπο να παρακάμπτουμε τους κανόνες που υπάρχουν και να φτιάχνουμε παραθυράκια να πετύχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε κάθε φορά. Άρα, το Συμβούλιο προφανώς χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια και ζητώ από την Προεδρία να κάνει ό,τι μπορεί για να το πετύχει αυτό και θα γίνει κλεισμένον των θυρών ε, μια συνάντηση με την Επιτροπή της Ομάδας Εργασίας για το ΣΕΓΕΝ. Ελπίζω να δημιουργήσει μεγαλύτερη σαφήνεια αυτό το πράγμα. Η κυρία Βερζιά θα θέλει το λόγο συντομία να απαντήσω γιατί η Γαλλία, να μου απαντήσετε στην ερώτηση γιατί η Γαλλία δεν περιλαμβάνεται στο, στην νομοθεσία αυτή. Η Επιτροπή θέλει να απαντήσει. Η Γαλλία είναι άλλη περίπτωση, διότι όπως αναφέρθηκε η Γαλλία για άλλη διαφορά παρέτεινε για σκοπούς αντιμετώπισης της τρομοκρατίας του έλεγχου στα σύνορα. Για τις άλλες πέντε χώρες οι λόγοι ήταν η μετανάστευση. Για την Ελλάδα και για την οδό των Δυτικών Βαλκανίων. Η Επιτροπή κοιτάζει και τις πιο πρόσφατες πληροφορίες της γαλλικής πλευράς για το θέμα αυτό. Άρα διαφορετικά σημεία του κώδικα Σέγγεν, διαφορετικά νομικά κριτήρια της ουσίας. Αυτή ήταν η τεχνική σας απάντηση. Συνοψίζοντας και χωρίς να ξεχνάμε πόσο σαφής ήταν ο κ. Κοέλιο στα τελευταία σχολεία του, να πω εγώ και να ενθαρρύνω την Προεδρία του Συμβουλίου να συντάξει σύντομα τις εκθέσεις του για να έχουμε τις σχετικές πληροφορίες διότι κανένα ζήτημα δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη πολιτική σημασία από αυτό. Και ε, καλό να είναι να έχουμε τις πληροφορίες αυτές για να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία του Σέγγεν και του θεσμού του. Αυτό δεν θέλουμε να χαθεί. Κάντε ό,τι μπορείτε λοιπόν. Και θα παρακολουθήσουμε στενά το θέμα. Καθώ και όσα είπε ο κύριο Κοέλιο για μια ενδεχόμενη και κλεισμένη των θυρών συνεδρίαση για να ενημερωθούμε καλύτερα για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέλιο και όλου του συναδέλφου που πήραν μέρο στην σχετική συζήτηση. Να είμαι τώρα στο σημείο 5 που είναι πρόταση για κανονισμό ε, για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της ενωσης Κανονισμό Κανονισμός 45-2001, κατάργηση αυτού δηλαδή, έκθεση της Κορνίλια Ένστ. Να περάσουμε στην παρουσίαση της έκθεσης από την Κορνιλία. Θα μας παρουσιάσετε σήμερα το σχέδιο έκθεσης. και μετά θα ακούσουμε και ε, τους εκπροσώπους της CDPS και ούτω καθεξής. Κορνίλια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλόντ. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω του σκιώτες που ήταν πάρα πολύ δραστήριοι στα πρώτα βήματα και στις συνεδριάσεις μας και την γραμματεία της ΛΥΜΠΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έδωσε πολλές πληροφορίες για τα σημαντικά ζητήματα της έκθεσής μας. Νομίζω ότι αυτά προκύπτουν και από την κοινή μας συζήτηση. Ένα σημείο θεωρώ ήταν αυτό στο οποίο είμαστε βέβαιοι και συμφωνούμε. Η εφαρμογή του βασικού κανονισμού για την προστασία των, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι τροπολογίε οι οποίε στο πλαίσιο αυτό Αυτό αφορά λοιπόν την εισαγωγή, την ε, δυνατότητα εισαγωγή ε, ε, πιστοποίηση για τι ευρωπαϊκέ υπηρεσίε και το θέμα που αφορούν το προσωπικό της γραμματείας. Αυτά είναι κάποια στιγμή τα οποία τα δουλέψαμε λίγο. Το βασικό ζήτημα στις συζητήσεις μας ήταν το θέμα του πεδίου εφαρμογή. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ συμφωνούν ότι για τον κανονισμό αυτό θα πρέπει να ισχύει όλη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι Πρόκειται δηλαδή για όρους που πραγματικά θα περιληφθούν στην έκθεση. Αυτό αφορά και τις υπηρεσίες, τις εξωτερικές υπηρεσίες Europol, Eurojust επίσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει σχετική ρύθμιση και αποφασίσαμε να με τρέπαθη στάση, να πούμε δηλαδή ότι όπου υπάρχει ε, ίδιο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων μεταβατικά θα εξακολουθήσει να ισχύει, αλλά μόνο στο βαθμό που συνάδει με την οδηγία του 2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. τα άλλα δεν έχει νόημα να διατηρηθεί το εθνικό σύστημα. Αυτό θα πρέπει να είναι αρχή μα. Ε, μέσω πρόθεσμα, και αυτό το αναφέρουμε σε ένα άρθρο, θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή με τον κανονισμό. Ωστόσο, το τρίτο θέμα είναι οι εσωτερικοί κανόνε, οι οποίοι εμφανίζονται σε διάφορα επίπεδα. Πιστεύουμε ότι ο περιορισμός της εξάσκησης των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων ατόμων θα πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα όπως και στο GPDR, δηλαδή τα δικαιώματα των ε, ατόμων τα οποία αφορούν τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να ρυθμίζονται από την νομοθεσία, όχι από εσωτερικού κανόνε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να, το εισαγω... να παραμείνει αυτή η ρύθμιση. Γι' αυτό λοιπόν και διαγράφουμε και τη δυνατότητα να υπάρξει παράκαμψη της νομοθεσίας μέσω εσωτερικών κανονισμών και να ρυθμίζονται ad hoc χωρίς νομική βάση. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί απόλυτα λογική συνέπεια. Άλλη μία προσαρμογή στον GPDR είναι η τροπολογία 26 για την προσαρμογή της νομοθεσίας όπως ισχύει για τα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο. Τέταρτο σημείο. Θα πρέπει να υπάρξει ένα κεντρικό μήτρο το οποίο θα πρέπει να τηρείται από τα κρατημέλη. Δεν είναι κάτι επίσημο αυτό, αλλά μια μεγάλη ανακούφιση για DPO σε ό,τι αφορά τα DPS, όπω μα είπαν. Πέμπτο σημείο. Έχουμε τα τρία άρθρα για το e-privacy, για την ηλεκτρονική αυτή ιδιωτική σφαίρα. Αυτά τα συζητιούνται διαρκώ. Και θεωρούμε ότι η βασική αρχή θα πρέπει να είναι ότι η ηλεκτρονική ιδιωτική σφαίρα προφανώς ισχύει και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αντίστοιχα θα ζητήσουμε κάτι τέτοιο με τροπολογίε για το e-privacy. Γι' αυτό έχουμε προσθέσει το άρθρο 35, γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό σε ό,τι αφορά την οδηγία για το e-privacy. Τα άλλα δύο θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Τώρα, έχουμε επανεισαγάγει το παλιό άρθρο 7. Αυτό μας το πρότεινε και ο EDPS, το οποίο ουσιαστικά υποχρεώνει να τηρηθούν όλοι οι νομοθεσίες σε ό,τι αφορά την φύλαξη δεδομένων από τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η υπεύθυνη επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο είναι απαραίτητη μεταφορά στοιχείων ή όχι. Και ένα δεύτερο θέμα είναι ότι κατά πόσον η μεταφορά των δεδομένων αυτών εξυπηρετεί δημόσιο και κοινό συμφέρον και γι' αυτό λοιπόν ε, ε Το EDPS θα πρέπει να διορίζεται λίγο πολύ όπως διορίζεται σήμερα, αλλά θα πρέπει να αποτελεί κοινή απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Προσαρμόσαμε λοιπόν μετά τις ε, τελευταίες εμπειρίες μας με τον διορισμό του EDPS. 8. 8 ζήτημα Υπήρξε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ξέρουμε ότι και εδώ χρειάζεται ανεξάρτητη επίβλεψη των δεδομένων και γι' αυτό λοιπόν καταθέσαμε τροπολογίες και έγιναν συζητήσεις για κυρώσεις. Εμείς δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει παρέκκληση από τους άλλους τομείς, ότι ισχύει και αλλού για τις, παρεκλη... Ε, κυρώσεις θα ισχύει και εδώ και ακολουθούμε και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Κορνίλια. Πάμε στους κοιόδες εισηγητές. Ο κύριος Φως. Ο κύριος Φως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κορνίλια Έρνης που κατέβαλε τόσο μεγάλες προσπάθειες από κοινού με τους κοιόδες εισηγητές και μας έχει ενημερώσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση εδώ είναι επί της αρχής απαραίτητη. Το είχαμε πει και για τον κανονισμό, βασικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, ότι θα πρέπει να ενταχθούν και τα θεσμικά όργανα και η εξίσωση μεταξύ κανονισμού και οδηγία του περασμένου έτους που συμφωνήθηκε πέρσι. Αυτό που είναι προβληματικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ έχει αναλάβει σε μεγάλο βαθμό το GPDR αλλά όχι πάντα εκεί που έχει νόημα. Η συνέντευξη παιδιών, για παράδειγμα, που αναφέρεται, αναρωτιέμαι. Μήπως είναι κάπως υπερβολικό αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπήρξε ενδελεχής εξέταση πριν τη μεταφορά και αυτό ισχύει και για τους ορισμούς. Αν θέλουμε να υπάρχει ένα ε, συνεκτικό σύστημα. Αυτό που είναι σημαντικό και ένα ερώτημα που θέλω να απευθύνω προς την εισηγήτρια είναι το εξή. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα σωστό εδώ σε θέματα ποινική συνεργασία και δικαστική συνεργασία και αστυνομική συνεργασία το πεδίο εφαρμογή τη πρόταση να διαφοροποιηθεί. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό εννοείται στην τροπολογία υπαριθμών 1, θέλουμε πραγματικά εδώ να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ε, λειτουργικών ε, και διοικητικών δεδομένων. Αν αυτό εννοείται, συμφωνώ και θα το υποστηρίξω. Για την τροπολογία υπαριθμών 5. Εδώ δεν νομίζω ότι καταλαβαίνω απόλυτα κατά πόσο να ε, θα απαγορευτεί η επεξεργασία η απαγόρευση επεξεργασία σε οποιοδήποτε ατόμων στην τροπολογία περιθμών 2 τώρα. Η εξίσωση με την οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φαίνεται ότι αφαιρέθηκε τι γίνεται και με τις εξωτερικές υπηρεσίε την Eurojust, την Europol, την ΕΠΟ, που έχουν ειδικό και χρειάζονται ειδικό καθεστώ για τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να κάνουν τη δουλειά του. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που ρωτώ είναι τα διοικητικά δεδομένα των ε, εξωτερικών αυτών υπηρεσιών να μην περιλαμβάνονται, αλλά τα λειτουργικά δεδομένα να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογή. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ. Αν αυτό εννοείται, σίγουρα θα το υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστέ, σοσιαλιστές παρακαλώ και όλες οι Η Μάριον. Ευχαριστώ την Κορνίγλια για την πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά της, για τις πολλές πληροφορίες που μας έδωσε κατά τη διάρκεια της σύνταξης της έκθεσης. Χαιρόμαστε που η Κομισιόν ε, ετοίμασε αυτή την έκθεση και μπορούμε να ολοκληρώσουμε το πακέτο για την προστασία των δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνει εδώ και τα θεσμικά όργανα. Βεβαίω, ο Ευρωπαίο Επόπτη Προστασία Δεδομένων ήταν το, η βάση του πλαισίου. μάθα που δεν εξετάσαμε και την ε, αστυνομική οδηγία. Ε, το, ήταν σημαντικό ότι εξετάσαμε τον κανονισμό, αλλά θα έπρεπε να δούμε και την οδηγία. Παραδείγματο χάρη τη μεταβίβαση των δεδομένων ή τον περιορισμό των ε, δικαιωμάτων ε, κατά τη διάρκεια τη δίκη. Ε, θα πρέπει να ξαναδούμε την οδηγία, την αστυνομική οδηγία. Αυτή η μειωμένη προσέγγιση, η μετριοπαθής προσέγγιση, μας επιβλήθηκε. Λόγω του ότι υπάρχουν ε, διαφορές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαιτίας αυτής της μετριοπαθούς προσέγγισης παραμένουν αυτές οι διαφορές. Στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε την, ε, το εγχείρημα αυτό, ακούστηκαν ιδέες ότι πιο σωστό θα ήταν όλο το σύστημα να επανεξεταστεί. Και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο, πραγματικά ενιαίο σύστημα. Συμφωνώ με την Κορνίλια, επίσης, για το θέμα των εσωτερικών κανόνων. Η αναφορά στους εσωτερικούς κανόνες, όταν μιλάμε για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των κατόχων των δεδομένων, ε, αν γίνει θα πρέπει να γίνει με τη σωστή νομική βάση. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά ακόμα, παραγωγική δουλειά. Και χαίρομαι που παράλληλα ε, κάναμε και τη δουλειά πάνω στο καονισμό για την ιδιωτικότητα, για την ιδιωτική σφαίρα. Ε, υπάρχουν αντιστοιχίες ε, και πρέπει βεβαίως αυτή η δουλειά να γίνει εκ παραλλήλου. Ο Ιαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια. Πάνω σε αυτή τη δουλειά, για αυτή τη δουλειά που έκανε για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν αυτά τα πρότυπα και σε όλους τους φορείς, σε όλα τα θεσμικά όργανα, σε όλα τα ιδρύματα, οι υπηρεσίες ε, επίσης. Δεν θα πρέπει να είναι ένας χωριστός κόσμος, δηλαδή διάφορες ε, υπηρεσίες να εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες. Φυσικά μπορούν να υπάρχουν και επιπλέον κανόνες πέραν του κανονισμού. Όταν όμως δεν υπάρχουν επιπλέον ειδικοί κανόνες, θα πρέπει να ισχύει ο κανονισμός. Τελεία. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λιγάκι αυτό, αυτή την ευκαιρία για να εφαρμόσουμε τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Γιατί αν μιλάμε, Φερρυπίν, για την πρόταση διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι προϋπόθεση να έχουμε... Βλέπω ότι είναι σημαντικό να έχουμε και πραγματική εναρμόνιση ε, στην προστασία των δεδομένων στο βαθμό που ανταλλάσσουν ε, δεδομένα οι διάφορες υπηρεσίες και τα διάφορα συστήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να κάνουμε αυτή την νομοθετική αλλαγή και να πιέσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν, καθώς και οι διάφορες agencies να συμφωνήσουν επί μίας κοινής δέσμης κανόνων. Επίσης, δεν θα πρέπει να συνεχίσει η πρακτική χρήσης εσωτερικών κανόνων και να είναι αυτή η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων. Και αυτές οι υπηρεσίες, όπως περιμένω και από τις αρχές των κρατών μελών και από τις διοκτικές ε, αρχές, να υιοθετήσουν νόμους, κανόνες οι δικοί μας κανόνες θα πρέπει να είναι αντίστοιχοι με αυτούς των κρατών μελών. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να, έχουμε, να επιτρέψουμε στην κάθε υπηρεσία να έχει τους δικούς της εσωτερικούς κανόνες. Αυτά περιμένω να εργαστούμε επί των κανόνων και επί των συμβασμών, συμβαστικών τροπολογιών δηλαδή, αλλά νομίζω ότι ήδη το πράγμα κινείται προς, προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Πρόεδρε τώρα, κύριε Τσιλιπέρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και καλημέρα σε όλους. Δύο τμήματα οι μου. Ε, διαδικασία και ουσία. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να ε, εξέρω την εξαιρετική δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το τελικό κείμενο του Συμβουλίου και η πρόταση κειμένου του εισηγητή ουσιαστικά κάνει χειρουργική φύσεως τροπολογίες σε ό,τι αφορά και τον επερχόμενη τριμερή διάλογο. Όντω, μετά τι 10 Ιανουαρίου, όταν η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύτηκε, έγινε μια σειρά συναντήσεων εμπειρογνωμόνων. Όταν διαβάσαμε όλα τα άρθρα και δύο και τρει φορέ, η, η Προεδρία πέρασε το κείμενο στου ε, Συμβούλου για θέματα ιστορικής ασφάλεια και δικαιοσύνη. και μετά περάσαμε σε επίπεδο Κορεπέρ και από 3 Μαου 2017 τεχνικός πω το θέμα αυτό ολοκληρώθηκε και την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων στι 8 Ιουνίου οι Υπουργοί ενέκριναν το κείμενο. Δηλαδή από σήμερα το Συμβούλιο είναι έτοιμο να αντιπραγματευτεί με το Συμβούλιο, με το Κοινοβούλιο βάσει του κειμένου επί του οποίου έχουν συμφωνήσει οι υπουργοί μα. Επί τη ουσία, τέσσερα είναι τα βασικά τα ζητήματα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά θα επικεντρωθώ στα τέσσερα αυτά τα οποία έχουν ε, σε μεγάλο βαθμό συζητηθεί και από την εισηγητρία. Το θέμα του πεδίου εφαρμογή, EDPS και σχέσει EDP και ε, ορισμοί να ξεκινήσω με το πιο εύκολο. διοικητικά πρόστιμα. Το Συμβούλιο ακολουθούσε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά του ιστορικού κανονισμού από μια πρώτη ανάγνωση τη έκταση του εισηγητή. Όντω, φαίνεται να υπάρχει συμφωνία επί τη αρχή όπου και το Συμβούλιο και η Συγήτρια αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Να απογορευτεί δηλαδή η δυνατότητα να υπάρχει εσωτερικό κανονισμό κατά απόκληση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ενδεχομένω να χρειαστεί βέβαια κάποια τεχνική προσαρμογή σε ό,τι αφορά η DPS, η DP. Το Συμβούλιο δεν έχει ακολουθήσει απαραίτητα, μάλλον έχει κάνει κάποιε μικρέ αλλαγέ σε σχέση με την πρόσθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όμω οδηγεί στο τέταρτο και βασικό ζήτημα, το θέμα του πεδίου εφαρμογή. και το τι έχει κάνει η, η Προεδρία εδώ. Έχει, α, αν θέλετε, χτενίσει λίγο καλύτερα το, το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν δύο, δύο υποζητήματα, υποθέματα εδώ πεδίο εφαρμογή από τον πρώην τρίτο πυλώνα. Έχει γίνει αναφορά στην Europol, Eurojust, EPPO και το πεδίο εφαρμογή σε ό,τι αφορά τον πρώην δεύτερο πυλώνα τις εξωτερικές υπηρεσίες που ήταν που θα μπουν στον τέταρτο πυλώνα. Αυτά έκανα λοιπόν το Συμβούλιο τους τελευταίους 4,5 μήνες. Τα βασικά, οι βασικές αρχές ήταν η συνοχή και η αναρμόνιση στο βαθμό του δυνατού με το GPDR. Ε, να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 25 Μαΐου του 2018 θα τεθεί σε εφαρμογή το GPDR. Έχουμε λοιπόν αυτό το χρόνο μπροστά μας. Ε, το Συμβούλιο είναι σε θέση και είναι διδεθμένο να διαπραγματευτεί με το Κοινοβούλιο και καλό την εισηγήτρια και τους κοιόδης να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους προκειμένου να περάσουμε σε διαπραγματεύσει και να βρούμε την απαραίτητη συμφωνία προκειμένου μέχρι 25 Μαΐου 2018 και το θέμα του GPDR και ο κανονισμός που ρυθμίζει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες να τεθούν σε εφαρμογή εκ παραλλήλου την ίδια ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μίκοφ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές για αυτή την έκθεση. Όπως και ο συνάδελφος από το Συμβούλιο, από την Προεδρία του Συμβουλίου, και εγώ συμφωνώ ότι που υπάρχει σύμπνη απόψεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για το στόχο αυτού του κανονισμού και την ευθυγράμμιση με αυτόν τον τρόπο, ε, με τον επόπτη Προστασία δεδομένων, Ευρωπαίο Επόπτη προστασία Δεδομένων, ολοκληρώνουμε το, όλο το μηχανισμό. Επίσης είναι σημαντικό να τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός ταχύτατα την ίδια στιγμή ε, μαζί με την αστυνομική οδηγία και το EDPR. Τον κανονισμό δηλαδή για την προστασία των δεδομένων. Υπάρχουν διάφορα θέματα και παρότι συμφωνούμε επί της ουσίας, υπάρχουν κάποια ζητηματάκια τα οποία θεωρούμε λιγάκι προβληματικά εμείς από πλευράς Κομισιόν. Θα ήθελα να σας τονίσω κάποια από αυτά. Η Προεδρία μόλις ανέφερε το θέμα των εσωτερικών κανόνων και της τροπολογίας 28. Και αυτό συζητήθηκε και στο Συμβούλιο. Για το, ποιο, για το ποια είναι η σημασία και η χρησιμότητα αυτών των εσωτερικών κανόνων και γιατί δεν μπορούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι, οι υπηρεσίες να βασιστούν σε διοικητικά κείμενα απλώς και μόνο. Είναι γιατί αυτοί οι φορείς δεν έχουν στη διάθεσή τους τα ίδια εργαλεία με αυτά που έχει ένα κράτος μέλος στη διάθεσή του. Μπορούν να, δεν μπορούν να έχουν ας πούμε προεδρικά διατάγματα τα οποία εξισώνται με νομοθετήματα. Για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τα νομοθετικά κείμενα έχουν πολύ πιο περιορισμένη εμβέλεια και πεδίο. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου να κάνει μια προσπάθεια ούτως ώστε αυτοί οι εσωτερικοί κανόνες να έχουν ε, το ύψος και την ποιότητα των ε, νομοθετημάτων είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι σωστός, ο σωστός δρόμος για να προχωρήσουμε. Αλλιώς θα επηρεαζόταν πάρα πολύ η δουλειά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ευρωπαϊκών οργανισμών. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι η τροπολογία 47 για το άρθρο 42 για την διαβούλευση των υπευθύνων προστασίας των δεδομένων. Η πρότασή μας είναι να διευκρινίσει τους τρόπους διαβούλευσης ανάμεσα στον EDPS και EDPB και για τις ε, κατεξιόδηση πράξεις, για τις ε, εκτελεστικές πράξεις και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άτυπες διαβουλεύσεις του, Ευρωπαϊ... του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ε, με τις, α, ε, τους υπόλοιπους υπευθύνους δεν θα λάβει χώρα. Εδώ μιλάμε για την υποχρεωτική όμως, την επίσημη αν θέλετε διαβούλευση. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να βάλουμε κάποιες ε, διατάξεις ακριβίας χωρίς να τροποποιήσουμε, να θίξουμε την άτυπη διαβούλευση που είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για τη σχέση αυτών των υπευθύνων προστασίας δεδομένων. Τώρα, κάποιες επιφυλάξεις σε κάποια άλλα σημεία για την εισαγωγή της υποχρέωσης να τηρείται ένα κεντρικό αρχείο. Θα πρέπει να κρατήσουμε τη δυνατότητα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να έχουν ε, κάτι τέτοιο εφόσον το επιθυμούν, αλλά να μην καταστεί αυτό μια υποχρέωση. Για τις τροπολογίες 22, την τροπολογία 22, που συνδέεται με το άρθρο 9. Πιστεύουμε ότι είναι λογικό να απαιτήσουμε ο αποδέκτης να αποδείξει ότι πρέπει να γίνει αυτή η διαβίβαση δεδομένων. Ότι χρειάζεται αυτή η διαβίβαση δεδομένων και, δεν χρειάζεται, και όχι να βαραίνει αυτή η υποχρέωση τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς. Τέλος. Έγινε μια τροπολογία, ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούμε πλήρως ε, με τον ε, κανονισμό σε κάποια άρθρα, με τον EDPR, τον κανονισμό προστασίας δεδομένων. Γενικά προσπαθήσαμε να σεβαστούμε και να ευθυγραμμιστούμε με τον ε, κανονισμό αυτό, αλλά κρατήσαμε κάποιες διατάξεις λόγω του προηγούμενου κανονισμού του 45-2001 που ήταν πολύ πιο προστατευτικός απέναντι στους υποκειμένους των δεδομένων, στους κατόχους των δεδομένων. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η ευθυγράμμιση λέξη προς λέξη. Τέλος, για την πιστοποίηση. Δεν νομίζουμε ότι είναι σωστό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι φορείς και οι υπηρεσίες, ας πούμε, και οι οργανισμοί να χρησιμοποιούν την πιστοποίηση. Πιστεύουμε ότι οι ιδιωτικοί φορείς πρέπει να κάνουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό δεν κρατήσαμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει στη διάθεση δηλαδή, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των οργανισμών κάτι τέτοιο, η πιστοποίηση δηλαδή. Κλείνοντα, η επανεισαγωγή του άρθρου 7 μέσω της τροπολογίας 21 σε όλες τις παρασκευαστικέ ε, εργασίες με σκοπό την κατάρτιση της ε, πρότασής μας δεν συγκεντρώσαμε αρκετά στοιχεία ε, υπέρ του άρθρου αυτού υπέρ της διατήρησης του άρθρου αυτού. Αντίθετα, προέκυψε ότι δημιουργεί πάρα πολύ σύγχυση στους εμπλεκόμενους. Γι' αυτό λοιπόν κρατήσαμε κάποια στοιχεία αυτού του παλιού άρθρου 7 σε μία στις αιτιολογικές σκέψεις, αλλά διαγράψαμε το άρθρο 7 από το διατακτικό του κειμένου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you. I'm going to return to Cornelia for πούμε και να δώσουμε το λόγο στην Κορνίλια για να κάνει τα καταληκτικά τη σχόλια, το επιθυμεί. Ναι, καταρχά σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλε αυτέ τι υποδείξει και τι δηλώσει mm. Ναι. από πλευρά των πολιτικών ομάδων και από την ε, Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το GPDR. Θα πρέπει να δούμε τι θα περιληφθεί και τι δεν θα συμπεριληφθεί. Χρειαζόμαστε διάκριση σε κεφάλαια, τι εννοεί εδώ το EPP Όλα αυτά θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε από κοινού. Αλλά δεν είδαμε σε πρώτη φάση κάποιο λόγο για να εξαιρεθούν κάποια κομμάτια για τα διοικητικά δεδομένα. Όχι, δεν θέλουμε να αφαιρεθούν. Όχι, ακριβώς αυτό είναι το θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει σε διάφορες περιστάσεις στις συναντήσεις μας. Δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση αυτό. Αν υπάρχει παρανάωση, μάλλον αν υπάρξει, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα το ξανακοιτάξουμε ενδεχομένω για το κατά πόσο δεν έχει λεφτεί υπόψη ε, επαρκώ η οδηγία. Να το κοιτάξουμε από πλευρά ε, σοσιαλδημοκρατών αν υπάρχει αυτό το θέμα. Όταν θα λάβουμε τι τροπολογίε, θα το εξετάσουμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά εναρμόνιση που θα αφορά και όλου του τομεί. Το παιδί εφαρμογή. Το πεδίο εφαρμογή ε, είναι ασφαλώ το πιο αμφιλεγόμενο σημείο. Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε το τι είναι το πιο ενδεδειγμένο, αν υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα Προστασία δεδομένων. Τι θα το κάνουμε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση σε κάθε περίπτωση και γι' αυτό λοιπόν κάναμε αυτή την πρόταση της συμβαστική στην τελική ανάλυση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτό το επόμενο βήμα. Ότι αυτό αναμένουμε. Το πρώτο βήμα λοιπόν θα αποτελέσει αυτό για να προσαρμοστούν τα συστήματα προστασίας δεδομένων με την οδηγία. Στο άρθρο 72α αναφέρουμε ότι θα πρέπει να αλλάξουν ενδεχομένως τα νομοθετικά, ή νομοθετικές διατάξεις. Αλλά αν υπάρχουν ε, άλλες προτάσεις, ε, με χαρά να τις ακούσουμε. Αυτή ήταν η δική μας πρόταση για το Μητρό. Είναι μικρή αυτή η πρόταση, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να έχει μεγάλα ωφέλη και να δίνει μεγάλες ε, δυνατότητες ε, συνολικής εποπτείας στους ε, επόπτες. Και αυτό μας το επεσήμαναν σε διάφορες περιστάσεις οι επόπτες. Το άρθρο 9 Μπορούμε θέλετε, να το ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό, γιατί εδώ το θέμα είναι η πρόσβαση στα δεδομένα και το πώς ε, όλοι μπορούμε να τα διευκρινίσουμε αυτά. Είναι αμφιλεγόμενο αυτό το διατυπώσαμε με μεγάλη προσοχή, αλλά μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε αν θέλετε. Εμείς θα θέλαμε να παραμείνει αυτή η διατύπωση, γιατί η πιστοποίηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είσαστε επικριτικοί. Εντάξει λοιπόν, να το ξανασυζητήσουμε αν είναι έτσι τα πράγματα. Εμεί θεωρήσαμε ότι αποτελούσε αυτό καλή προσθήκη και μία λύση από πλευρά του GPDR την οποία θα θέλαμε να επιτηρήσουμε. Αυτά ίσως επί του παρόντος για τους ιστορικούς κανόνες. Εδώ πραγματικά δεν υπάρχει μεγάλη, μεγάλο πάθος. Θέλουμε να παραμείνουμε στη γραμμή μας. Γιατί για μας δεν υπάρχει κανένας πραγματικός λόγος για όλα αυτά που τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε να γίνουν γρήγορα οι διαπραγματεύσει για την τη συμβιβασμού. Ελπίζουμε λοιπόν να είναι γρήγορη η διαδικασία και νομίζω ότι είμαστε ακόμα μέσα στα χρονικά περιθώρια τα οποία προβλέπονται. Σα ευχαριστώ, Κορνελία, Ευχαριστώ και του Κιώδη. Και την ε, Προεδρία και την Επιτροπή. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 11 Ιουλίου στι 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. We move now to the... Περνάμε τώρα στο σημείο 6 ή privacy. Η πρόταση για την ε, ηλεκτρονική προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση που θα ε, συμπληρώσει τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ξεκίνησε με την μεταρρύθμιση του GDPR το 2016. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και η Συγγήτρια Όλος Ιδιαίτερος έχουν εργαστεί εντατικά τις τελευταίες εβδομάδες και σήμερα θα περάσουμε στην παρουσίαση της έκθεσης της Μαριού Λάουριστην Μαριού, να σου δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσή σου. Παρακαλώ, πάρε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για αυτή την ε, ευκαιρία. Και εγώ να εκφράσω τις βαθιές μου ευχαριστίες προς όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, αυτή την εντατική διαδικασία σύνταξη της έκθεσης, ξεκινώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άριστη συνεργασία που είχαμε για το άρθρο 29 που φέρνει επιτάκτως πολλές σημαντικές ιδέες, όλους τους σκιώδεις και τους βοηθούς τους που συμμετείχαν στις συζητήσεις μας με τους ενδιαφερομένους, ε, συζητήσεις τρογγυλής τράπεζας και βεβαίως τους συνεργάτες και βοηθούς μας, την Ελένη, τη και όλους τους υπόλοιπους που συνέβαλαν στην σύνταξη της έκθεσης αυτής. Ελπίζω πραγματικά ότι καταλήξαμε σε μια καλύτερη και πιο ευρεία κατανόηση όλων των θεμάτων που θα απασχολούν εδώ. Ε, το σημείο αφετηρίας που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ή ήταν πολύ καλό. Όμως τις συζητήσεις που είχαμε μεταξύ μας και με τους ενδιαφερόμενους προσπαθήσαμε να δούμε θέματα που παραμένουν κάπως αμφιλεγόμενα, όπου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Τα θέματα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με, για τη της, ε, προς τη σχέση του κανονισμού GDPR, ε, όπως λέει ονομαστεί, και του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η οδηγία δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις επικοινωνίας δεν καλύπτει αυτά που συμβαίνουν με την σύγκληση των μέσων μαζική ενημέρωση, με όσα έχουν ε, γίνει με το ξέσπασμα και την, ε, την τεράστια άνθηση των ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή της διασύνδεσης των συσκευών. Από την άλλη, ο κανονισμός GDPR έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό και ισχυρό πλαίσιο, γενικό πλαίσιο και αυτό είναι και το ερώτημα. Πού είναι οι διαφορές και που οι κανονισμοί για την ηλεκτρονική ε, ιδιωτικότητα ε, είναι, ε, κινούνται σε άλλους τομείς ή επικαλύπτουν τον κανονισμό GDPR. Το πρώτο και πλέον σημαντικό που να θυμόμαστε είναι ότι ο κανονισμός GDPR βασίζεται στο άρθρο 8 της Σύμβασης για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για την προστασία των δεδομένων, ενώ ο κανονισμός e-privacy βασίζεται στο άρθρο 7 προστασία του απορρίτου και της εμπιστευτικότητας του ιδιωτικού βίου. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και δεδομένων. Πολύ περίπλοκο βέβαια, γιατί έτσι είναι και το θέμα του ιδιωτικού βίου αυτό καθεαυτό. Η προστασία του ιδιωτικού βίου λοιπόν δεν είναι ε, δικαίωμα ε, από καιρού εις καιρών. Μιλάμε για την προστασία της ατομικότητας, την ε, ελευθερία συνείδησης, έκφρασης, όλα αυτά τα στοιχεία. Άρα είναι κάτι το πολύ βασικό και θεμελιώδες. Και η εμπειρία μας ως τώρα από τα διάφορα συστήματα είναι ότι ο ιδιωτικός βίος είναι το πλέον σημαντικό ε, στοιχείο, γιατί εφόσον αποστερηθεί αυτό δεν υπάρχει καμία άλλη αίσθηση ελευθερίας στους ανθρώπους. Τώρα, ως προς το πεδίο, υπάρχει και εκεί κάποια, ε, κάποιος διότι το βασικό σημείο είναι τι συμπεριλαμβάνουμε όταν μιλάμε για ηλεκτρονική επικοινωνία και αν ε, εννοείται και επικοινωνία μηχανής προς μηχανή, συσκευής προς συσκευή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ορισμό τη λέει κάτι το κάπως ασαφές, ε, δεν ήταν σαφές που είναι το όριο δεν ήταν σαφές εάν η μηχανή προς μηχανή επικοινωνία καλύπτεται εάν τα ανθρώπινα όντα ε, που ε, εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς ε, εδώ καλύπτονται. Έπρεπε λοιπόν να αποσαφηνίσουν τον ορισμό λέγοντας ότι στο πεδίο δεν, δεν, στο πεδίο δεν περιλαμβάνονται όλες οι από μηχανή προς μηχανή επικοινωνίες αλλά μόνο όταν συμπεριλαμβάνεται και άνθρωπος, άτομο στις μηχανές αυτές στις συσκευές. Άρα μπορεί να μην έχουν σχέση με τα προσωπικά δεδομένα αυτές οι διασυνδέσεις. Κάτι άλλο που παραμένει επίσης συζήτηση είναι οι επικουρικές υπηρεσίες που σχετίζονται με άλλες υπηρεσίες. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα ιδιωτικότητας, ιδιωτικού βίου. Και πρέπει και αυτά να καλύπτονται. Αν προχωρήσουμε τώρα με το πεδίο, σημαντικό είναι να δούμε όχι μόνο την επεξεργασία των πληροφοριών, δηλαδή τη μεταφορά πληροφοριών, αλλά και το τερματικό που χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός. Διότι αν δείτε τις δυνατότητες που έχουν πλέον οι συσκευές, ας πούμε τα smartphone, η δυνατότητα αποθήκευσης ε, των εξοπλισμών αυτών αυξάνεται καθημερινά. Είναι απίστευτος ο αριθμός δεδομένων που μπορεί να διαθέτουν για τη ζωή μας, για τις επαφές μας, για κάθε φάση της δραστηριότητάς μας. Ο εξοπλισμός λοιπόν αυτός, η συσκευή αυτή, είναι και αυτή μέρος του ειδητικού βίου. Έτσι, το πεδίο χρησιμοποιείται τερματικά, τις συσκευές και τα αρχεία που τηρούν και το πώ επεξεργάζονται τις πληροφορίες. Έπειτα, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνονταν όχι μόνο τα άτομα και τα πρόσωπα, τα φυσικά, αλλά και τα νομικά. Αυτό δημιούργησε κάποια σύγχυση. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδιωτικό βίο νομικών ε, προσώπων. Διότι αυτό μπερδεύεται μετά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Υπήρχε το πρόβλημα λοιπόν τη ε, εμπιστευτικότητα και του απορρίτου στην επικοινωνία με τα νομικά πρέσια και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε το διαχωρισμό στον ορισμό χρησιμοποιούσαμε δύο διαφορετικούς όρους, το χρήστη και τον τελικό χρήστη. Ο τελικός χρήστης είναι ε, φυσικό πρόσωπο. Όταν ε, ε, μιλάμε για χρήστη γενικότερα μπορεί να εννοείται και νομικό πρόσωπο. Πολλά άρθρα λοιπόν κάνουν λόγο για χρήστη και εννοούν ακριβώς τα νομικά πρόσωπα. Τώρα, το άλλο πρόβλημα είναι ότι ο κώδικα των τηλεπικοινωνιών δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει περατεθεί. Εδώ λοιπόν υπήρχε ένα ζήτημα. Ε, ε, στην αρχή είχαμε μόνο παραπομπέ στο κείμενο τη Επιτροπή. Το ανοίξαμε και αυτό το θέμα και κοιτάξαμε να συμπεριληφθεί ακριβώ το κείμενο όπω είναι στον κώδικα με κάποιε τροποποιήσει. Και όταν τελικά θα έχουμε έτοιμο τον κώδικα και θα έχει περατωθεί, θα φροντίσουμε να υπάρξει απαραίτητη αντιστοίχηση. Έπειτα σημαντικό είναι Α, σημαντικό είναι να πούμε ότι το άρθρο 5 τώρα έχει διατυπωθεί ως μια κεντρική σημασία δήλωση για όλο τον κανονισμό. Για τις τηλεπικοινωνίες, τον ε, εξοπλισμό και τις θερματικές συσκευές, και ξεκαθαρίζει τα όρια του πεδίου. Ε, ε από αυτό το άρθρο ε, εκπορεύονται και κάποιες ε, προϋποθέσεις. Η εμπιστευτικότητα, το απόρριτο, που επιτρέπει κάποιες εξαιρέσεις. Στο κείμενο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη υπήρχαν τα στοιχεία αυτά, αλλά προσπαθήσαμε να τα αποσαφηνίσουμε, να τα παριθμίσουμε πιο καταλεπτός, διότι οι συζητήσει με του ενδιαφερομένου για το GDPR, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεν μπορεί να εννοεί εδώ το γενικό δικαίωμα για την παραβίαση του ιδιωτικού βίου. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ διεξοδική απαρίθμηση, ώστε να είναι σαφές που η επεξεργασία των δεδομένων είναι νόμιμη ή όχι. Ως προς τις τηλεπικοινωνίες αλλά και τον ε, εξοπλισμό τερματικού μια από τις μείζονε αλλαγέ η καινοτομίες αν θέλετε του κανονισμού αυτό, αυτό που προσπαθήσαμε να προσφέρουμε εμεί είναι η δυνατότητα του χρήστη να προστατεύσει την ίδια την ιδιωτική του ζωή. Διότι ενώ ευρέω αναγνωρίζετε ότι το βασικό θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν κατανοεί και δεν χρησιμοποιεί όλες τις ευκαιρίες που έχει αυτές που προσφέρει η τεχνολογία για να προστατεύσει τον ιδιωτικό του βίο, από άγνοια δεν καταφέρνει να κάνει τις σωστές ρυθμίσεις λόγου χάρη. Και πολλές φορές και οι πάροχοι αντιστρέφουν την ευθύνη και τη φορτώνουν στο χρήστη. Και τους λένε, μπορείτε, λένε στο χρήστη μπορείς να κάνεις opt-out, να εξαιρεθείς. Τώρα με την ενιαία ψηφιακή αγορά, ε, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι με τα παιδιά, οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι ηλικιωμένοι, μπορεί να χρησιμοποιούν τεχνολογία και τεχνολογικά μέσα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχουν επίγνωση και ευθύνη για το πώ θα χρησιμοποιούν αυτές τι περίπλοκες διαδικασίε στι συσκευέ του. Προτείνουμε λοιπόν οι αρχικέ ρυθμίσει. να είναι αυτό που ε, ονομάζουμε donor track. Δηλαδή, ο χρήστης να έχει ήδη τις σωστές ρυθμίσεις και όταν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή να λαμβάνει γνώση για την αλλαγή. Κάτι που ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο σε σχέση με το κείμενο της Επιτροπής ήταν τα cookies ε, ε, από τρίτα μέρη. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε τα cookies. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της καταγραφής στοιχείων και μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο χρήσιμα, παρεμβατικά και ούτω καθεξής. Πάντως χρησιμοποιούνται εργαλεία ε, καταγραφής μιας διαδρομής. Προσπαθήσαμε λοιπόν να μην κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ πρώτων και τρίτων μερών και ακολουθήσαμε μια προσέγγιση πάρα πολύ ε, διεξοδική, λεπτομερή. Ως προς το GDPR, τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, κοιτάξαμε τι είναι ο ιδιωτικός βίος by default και by design, δηλαδή καταρχήν και βάση ρυθμισής, ε, ε, του σχεδιασμού Ο σχεδιασμός υπονοεί ότι οι Ευρωπαίοι πάροχοι και σχεδιαστές μπορούν να αναπτύξουν νέα τεχνολογικά μέσα για να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εφόσον επιζητούν λύσεις σε αυτά τα τόσο περίπλοκα ζητήματα. Αυτό που είναι πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες που συναντήσαμε εκπροσώπους τους, συναντήσαμε ε, ενδιαφερομένους από διάφορες εταιρείε και πολλές εταιρείε έχουν προτείνει ε, την ε, λύσεις για την διαχείριση της ιδιωτικότητα. Στη Μάλτα πρόσφατα είχαμε μια διάσκεψη για τις νέες τεχνολογίες λόγω χάρη και ήταν φοβερό πώ οι εταιρείε έρχονταν να μας παρουσιάσουν για την προσέγγιση αυτή ακριβώ νέε λύσει. Ελπίζω λοιπόν ότι εδώ θα δώσουμε μια όθηση προς την ανάπτυξη ευρωπαϊκών λύσεων. Τώρα, η θεσμική πλευρά. Η θεσμική πλευρά της παρακολούθησης του ελέγχου και ούτω καθεξής έχει ευθυγραμμιστεί με την προστασία των δεδομένων οι ίδιε αρχέ έχουν αναλάβει αυτά τα καθήκοντα και το Συμβούλιο Προστασία των Δεδομένων ε, παρακολουθείται και από εμά και ασχολείται με πολλά περιπλοκά ζητήματα. γιατί τη λόγου χάρη, έναν αναφέρω, ύψη τη σημασία πώ να προστατεύονται καλύτερα τα παιδιά. Προσπαθήσαμε να βρούμε λύσει και ακόμη αναζητούμε τι καλύτερε, αλλά είναι πολλέ λεπτομέρειε που πρέπει να αποσαφανιστούν. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο Λόγου Προστασία Δεδομένων θα διευκολύνει και τη δουλειά των παρόχων. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνοχή μεταξύ του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων και του κανονισμού για την προστασία του ιδιωτικού βίου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε την ίδια περίοδο υλοποίηση. Χθες, η κυρία Γκάμπριελ που απαντούσε στις ερωτήσεις μας, το τόνισε και χάρηκα πολύ που το άκουσα, αλλά είπε ότι η προτεραιότητά μας και για τους δύο κανονισμούς είναι να προχωρήσουν παράλληλα, να συμβαδίσουν, για να υπάρχει και θεσμική συνέπεια, να μην δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ χρηστών. Προτείνουμε, όπως εργαζόμαστε βάσει αυτού του αυστηρού χρονοδιαγράμματος, Ε, προτείνουμε να και επιδιώκουμε να έχουμε ολοκληρώσει στο φθινόπωρο. Τι τροπολογίε θα θέλαμε να τι λάβουμε πριν την καλοκαιρινή διακοπή για να τι επεξεργαστούμε κατά τη διάρκεια των διακοπών και να τι έχουμε έτοιμε μέχρι το τέλο ε, των διακοπών το Σεπτέμβριο. Τελευταία λοιπόν ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 10 Ιουλίου στις 3, ενώ πριν λέγαμε 5. 10 Ιουλίου στις 15.00 ε, παρακαλώ στείλτε μας τις τροπολογίες σας. Σας ευχαριστούμε. Πάντα η παρουσίασή σας είναι ενθουσιώδης. Λες και η πρώτη φορά που κάνεις παρουσίαση. Να σας πω ότι η ψηφοφορία είναι στις 12. Ξέρω ότι θέλω να πάρω το λόγο και οι Αλλά σας παρακαλώ να είστε συνοπτικοί. Να σας διαβάσετε τον κατάλογο, αν δεν θέλει κανένας άλλος. Is there anyone else that wants... Άλλος κανείς που θα θέλει να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Αν όχι, να κλείσω τον κατάλογο και να σας πω ότι έχουμε μέχρι τις 12. Κύριε Μπούνη. καταρχάς. Thank you very much. Ε, ε. Σας ευχαριστώ. Και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίαση της έκθεσης αλλά και για την καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της έκθεσης. διοργανώθηκαν ε, στρόγγυλες τράπεζες με εκπροσώπους ε, των ενδιαφερομένων. Αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο και έτσι κατανοούμε πολύ καλύτερα την ε, κατάσταση. Ο στόχος αυτή του κανονισμού είναι να βελτιώσει την αξιοπιστία και την ασφάλεια των επικοινωνιών. Σύμφωνα με αυτά που είπε η Μαριού, ότι η βάση δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τα δεδομένα, αλλά με την ιδιωτική ζωή και όλη την έκφραση και την έκφανση, αν θέλετε, τη ιδιωτική ζωή. Κατανοούμε λοιπόν την ανάγκη να ενημερωθούν όλα αυτά τα δεδομένα των τεχνολογικών εξελίξεων, να μην ξεχνάμε τον άλλο στόχο. Την ελεύθερη ροή δεδομένων. Αυτό δεν σημαίνει μόνο προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικότητα, θα πρέπει να το θυμόμαστε όμως σίγουρα πάντα αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνο ότι σκοπός είναι της πρότασης να εγγυηθούμε πραγματικά το απόρριτο της ε, επικοινωνίας και άρα θα πρέπει αυτό να ισχύει για όλους τους παραόχους ε, ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει να καλύπτεται, αλλά το πώς θα πρέπει να καλύπτεται να σκεφτούμε κάποιες ε, ισορροπημένες λύσεις ε, στις τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να ενισχύσω την εξέριξη και την ασφάλεια στην πρόταση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό για την ασφάλεια όλων των χρηστών και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι λύσεις μας είναι συνοπτικές, συνεκτικές με τον κώδικα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν Μάριον που είσαι πρόθυμη να προσαρμόσεις τον ορισμό σε όσα έχουν ε, καταλήξει και από το πλευρά του Συμβουλίου. Και επίσης ότι θα πρέπει να πετύχουμε εναρμόνιση με τον GPDR προκειμένου να μην υπάρχουν αντιφάσεις. Αναφέρατε και αυτό περιλαμβάνεται και στο σχέδιο έκθεσή σας άλλωστε κάποιες επιπρόσθετες λύσεις σε ό,τι αφορά την M2M, machine to machine. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο από πλευρά τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ είμαι διστακτικό. Πρόκειται για μία ιδέα και μόνο. Δεν είμαι βέβαιο μήπω είναι υπερβολικά νωρί να τα περιγράψουμε αυτά, αλλά θα εξετάσω τι ε, λύσει που προτείνονται και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι λύσει που εφαρμόζουμε θα είναι τεχνολογικώς ουδέτερες και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία στην όλη αυτή διαδικασία, σε όλη αυτή την πρόταση. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα browsers και τα cookies, όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι κόβουλα όλα τα cookies τρίτων μερών. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε το στόχο τους και να εξασφαλίσουμε ότι ο τελικός χρήστης γνωρίζει το τι συμβαίνει με τα δεδομένα τους. Και θα είναι σε θέση να κάνει μια ενημερωμένη επιλογή και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κίνητρα για τις εταιρείε προκειμένου να δίνουν λύσεις φιλικές προς την προστασία των δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ενημέρωσης και της ε, πληροφόρησης ε, των ατόμων και των εταιριών που θα είναι πιο πρόθυμες να προβούν σε λύσεις που θα συνάδουν με, την, με το απόρριτο. Και επίσης σε ό,τι αφορά τα θέματα των καινοτομιών, τα big data, θα τα εξετάσω και τα θέματα προστασίας των δεδομένων. Καταλαβαίνω ότι μπορούμε να είμαστε πιο φιλοδοξοί για να επιτρέψουμε καινοτομία σε διάφορους τομείς για την προτέρα επεξεργασία των δεδομένων, ενώ παράλληλα ε, θα εισάγουμε τις απαραίτητες και αυστηρές ε, ε, δικλείδες ασφαλείας. Στο άρθρο 11 της πρότασης μιλάμε για περιορισμούς. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεπεράσουμε την δικαστική απόφαση, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. σε ό,τι αφορά την ευελιξία που θα έχουν δηλαδή τα κράτη-μέλη για να προσαρμόσουν την ομοθεσία. και τελικά να περάσουν σε, κάτω, σε κάτι το οποίο θα είναι κατά τη ε, προστασία των δεδομένων. Επίση, αναρωτιέμαι σε ό,τι αφορά την εφικτότητα του κανονισμού αυτού που θα τεθεί σε εφαρμογή χωρί ε, περίοδο μετάβαση για την προσαρμογή των εμπλεκομένων φορέων. Ιδιαίτερα αν απαιτήσουμε να εισαχθούν νέε τεχνικέ λύσει, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να εξετάσουμε κατά πόσον είναι εφικτή αυτή η λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να αναβληθεί η εργασία της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά στην τελική ανάλυση να δούμε και το πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Αναλύοντας την πρόταση σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας, είμαι βέβαιος ότι θα είναι εξαιρετική η συνεργασία μας και με την εισηγήτρια και με τους σκιώδεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μέχρι τις 10 Ιουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος από το ECR, σκιώδης ε, του ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια ε, για την διάθεση να μας ακούσει από την αρχή της διαδικασίας. Όμως έχω παρόλα αυτά σοβαρές ανησυχίες. Καταρχάς, με την πρόταση της Κομισιόν, ήδη από τότε ανησυχούσα. Όταν για το σχέδιο έκθεση, ας ανησυχώ ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι θα καταστεί η κατάσταση πολύ πιο δύσκολη για τα άτομα, για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές όλος ιδιαίτερος. Καταρχάς το χρονικό πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό αυτό το χρονικό πλαίσιο με βάση το οποίο δουλεύουμε. Καταρχάς μόλις συμφωνήσαμε τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, ε, ο οποίος δεν είναι ακόμα σε ισχύ. Νομίζω ότι πολύ πιο λογικό θα ήταν να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο κανονισμός, τι προβλήματα παρουσιάζει και συνεχεία ε, να το αντιμετωπίσουμε. Όταν τα είπα αυτά στην Επιτροπή, ο κ. Άλμπρεχτ μου είπε ότι δεν συνειδητοποιώ ότι έχουμε ένα κανονισμό για την ιδιωτική σφαίρα. Φυσικά και έχουμε, αλλά θα πρέπει να ανακληθεί ούτω ώστε να προχωρήσει ο καινούριο. Έχουμε προστασία τη ιδιωτική σφαίρα, ούτω ή άλλω. Ε, α περιμένουμε, α δούμε ποια προβλήματα θα προκύψουν με τον κανονισμό κατά την εφαρμογή του και συνεχεία να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό για την ιδιωτική σφαίρα. Αυτή θα ήταν μια πιο λογική προσέγγιση, καλύτερη νομοθετική διαδικασία. Όμω έχουμε την πρόταση τη Κομισιόν και ω Επιτροπή θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μα, να τη θεωρήσουμε. Παράλληλα, όμω, ε, ε, αναθεωρούμε και τον κώδικα επικοινωνιών. Παράλληλη διαδικασία. Ε, Επομένω, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε και με αυτό. Αλλιώ θα τα κάνουμε όλα μαντάρα, ειδικά στου ορισμού. Νομίζω ότι οι ορισμοί θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον κώδικα αν θέλουμε να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές να έχουν ε, νομική βεβαιότητα και κυρίως ε, για τις ε, δευτερογενείς υπηρεσίες, τις δευτερεύουσες υπηρεσίες, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη δυνατή μεταχείριση. Σε ό,τι αφορά την έκθεση, είναι πολύ στενή η προσέγγιση για την συνένεση με σκοπό την επεξεργασία. Είμαι κατά για δύο λόγους. Καταρχάς, είναι πάλι διαφορετικό από τον κανονισμό με τον οποίο μόλι συμφωνήσαμε και να έχει τεθεί καν σε εφαρμογή. Επομένω, πέστε μου, τι πρόβλημα έχει ο κανονισμό. Μόλι το συμφωνήσαμε. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι θαυμάσια η πρόταση. Προλίγου τα λέγανε αυτά και τώρα αρχίζουμε να παρεκκλίνουμε ήδη. Και δεύτερον, παρεκκλίνουμε από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κάτι που θεωρώ πάρα πολύ περίεργο, γιατί στο άρθρο 8 τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων λέει ξεκάθαρα ότι κάθε ένα έχει ε, δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων και αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να τυχάνουν επεξεργασία ε, για συγκεκριμένους λόγους και όχι βάση ε, της συνέντευξης των προσώπων. Γιατί κλείνουμε από την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε αυτόν τον τομέα. Ε, δεν είναι πρακτικό. Δεν, δεν δικαιολογείται ούτως ή άλλως. Όταν μιλάμε για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας επίσης, δεν καταλαβαίνω ε, τι σημαίνει αυτή η επικοινωνία μηχανή προς μηχανή, κυρίως σε ένα πλαίσιο ε, επιχειρηματικών ε, σχέσεων, σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Ε, θα το συζητήσουμε και μετά, αλλά νομίζω ότι είναι λογικό. Για ποια, ε, ποια ε, ιδιωτική ζωή μιλάμε. Εδώ μιλάμε για μηχανές, έτσι. Σε ό,τι αφορά τη συνένεση και τα cookies, επίσης ανησυχώ για τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζουμε. Νομίζω ο, ο browser ως φύλακας, ας πούμε, είναι λάθος προστασίας. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Και δεύτερον, ε, το να ζητάμε αυτή την συνένεση και μετά να ζητάμε συνένεση εκ νέου κάθε 6 μήνε, ε, θα υπάρξει μια κόπωση, ας πούμε, τη πολλαπλέ συνενέσει. Έλεω. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι θα υπάρξει τέτοια συγκέντρωση ας πούμε, δεδομένων που θα καταληθεί το μοντέλο του ίντερνετ όπως το ξέρουμε σήμερα, το οποίο λειτουργεί με βάση την διαφήμιση. Γι' αυτό ακριβώς η μεγάλη πλειοψηφία του ίντερνετ είναι ε, ελεύθερη. Ε, και όταν ε, δεν πληρώνεις, και όπου δεν πληρώνεις την πραγματικότητα, επιδοτείται από τις διαφημίσεις. αλλιώς, με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πολύ πιο... Θα, Παραδείγματο χάρη, αν απαγορεύσει τι διαφημίσει, θα πρέπει να πληρώνει παντού. Και καλά, ε, άμα είσαι ας πούμε πλούσιος κτλ. Αλλά τι θα γίνει με τους νέους που δεν έχουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ε, Ποιο θα πληρώσει, εν πάση περιπτώσει, μόνο και μόνο αν αυξήσουμε τι τιμέ, είναι γελίο. Και επιπλέον, α ξεκαθαρίσουμε ότι ο κόσμο ούτω ή άλλω επιλέγει σε όλα αυτά. Εάν ξέρει τι σημαίνει κούκι, ξέρει πολύ καλά πώ μπορεί να διαγράψει το κούκι από τον υπολογιστή σου. Εάν δεν ξέρει, ούτω ή άλλως ε, το δέχεσαι γιατί δεν ξέρει τι κάνει. Όλα τα μέτρα υπάρχουν σε όλου του υπολογιστέ, ούτω ώστε να μπορούμε να καλύψω, καλύπτουμε τα, τα ίχνη μας. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει ε, να τα καταλάβουμε όλα αυτά ε, και να καταλάβουμε πώ λειτουργεί το ίντερνετ πριν αρχίσουμε να χλεβάζουμε για το μέλλον. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Μπόνι για τι εξαιρέσει για την ασφάλεια. Είναι πολύ λογικό να το εξετάσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλε. Ε, ιδιωτικές ε, επιλογέ που να βασίζονται στην αγορά, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι τεράστιο νομοθετικό θέμα. Επηρεάζει τα πάντα, κάθε κλάδο, ε, κάθε οικονομική δραστηριότητα, κάθε άτομο και θα πρέπει να είμαστε σωστοί. Έχω θέσει διάφορε ανησυχίε και περιμένω να αντιμετωπιστούν, να εξεταστούν, να απαντηθούν. Επίση, θέλω να συνεργαστώ πολύ στενά με τους σκιώδεις εισηγητέ, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η συμφωνία τελικά είναι καλή. Αλλά υπάρχουν τεράστια προβλήματα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Πέρα από αυτό. Σα αρέσει όμως, ε. Α, ωραία, τέλεια, μπράβο. Ευτυχώς. Εντάξει, δεν θέλω να υποβαθμίσω τα επιχειρηματά σα. Α, τέλο πάντων, τελειώνουμε με έναν αναστεναγμό ανακούφιση. Α, ουφ. Για να καταλάβουμε όλοι τι ακούμε. Έτσι η Σόφη Ιντβελτ, σκιώδης των φιλελεύθερων. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να σα εξοικονομήσω χρόνο και να τα πω λακωνικά και να πω ε, τι ακούσατε να σας λέει αυτός, όλα ισχύουν από την αντίθετη όμως, από την ανάποδη. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κυρίως γιατί εξασφαλίζει ότι κάτι θα έχω να κάνω και το καλοκαίρι, έτσι αλλιώς θα βαριόμουν, θα σκυλοβαριόμουν. Ε, σας ευχαριστώ, χωρίς πλάκα τώρα, για μια πολύ καλή πρόταση που υποβάλλετε. Την έχετε σκεφτεί, την προετοιμάσατε πολύ ενδελεχώς, ε, έχετε μία ανοιχτή ε, προσέγγιση, ε, ακούσατε όλους τους εμπλεκόμενους και προσπαθήσατε να κάνετε προτάσεις οι οποίες να διασκεδάζουν όσο να τον περισσότερες ανησυχίες. Ένα πρόβλημα με το οποίο θα μπορούσα να είχα συμφωνήσει στο, στην ομιλία Ντόλτον είναι ότι επηρεάζει όλα τα άτομα, τους πάντες. Μα ε, περί αυτού πρόκειται, γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να προστατεύονται. Και Διαφωνώ θεμελιακά με αυτή τη δήλωση η οποία έχει παγιατέψει πια. Έτσι, τα ίδια και τα ίδια μας κοπανάτε εδώ πέρα. θα, διαλυθεί το ίντερνετ και θα καταρακωθούν οι επιχειρήσεις. Τα ακούμε χρόνια αυτά. Και το ίντερνετ είναι ζωντανό, Ζωντανό ζωντανότατο και αν υπάρχει πρόβλημα νομοθετικό, λογικό είναι γιατί νομοθετούμε για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Δεν είμαστε στη ζούγκλα, έτσι. Έχουμε νόμους και προστατεύουμε τους ανθρώπους και οι επιχειρήσεις ούτω ή άλλω βρίσκουν καινοτόμου τρόπους για να παρακάμπτουν τα εμπόδια. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να πετύχουμε εδώ. Δεν θα μπω τώρα σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί είναι κάτι εξόχως πολιτικό. Οι περισσότεροι από τους πολίτες μας ανησυχούν πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί θέλουν να χρησιμοποιούν το ίντερνετ, θέλουν να χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε του, να επικοινωνούν, αλλά φυσικά θέλουν να είναι σίγουροι ότι οι επικοινωνίε είναι ιδιωτικέ και ότι προστατεύονται. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα αυτό. Και ο κύριο Ντόλτον είπε ότι πάμε υπερβολικά γρήγορα, ότι κάνουμε fast forward και θα πρέπει να περιμένουμε. Το ίντερνετ δεν περιμένει. Όταν κάναμε την προηγούμενη αναθεώρηση τη ε, οδηγία για την ιδιωτική σφαίρα, δεν είχαμε το iPhone καν στην αγορά. Για να καταλάβετε πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα πράγματα. σα τα λέω αυτά. Είναι πολύ επίκαιρη λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Ένα τελικό σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα και καλωσορίζω το σχόλιο του Μιχαήλ Μπόνη για το άρθρο 11. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να γίνει αλλαγή. Στο παλιό, στο αρχικό άρθρο 15 δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι εκτός του πεδίου της αναθεώρησης ε, που έχει να κάνει με τις ε, τεχνολογικές εξέλιξεις. Και δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί θα πρέπει να διευρύνουμε περαιτέρω το επαρκώς ευρύ πεδίο που έχουν τα κράτη-μέλη για να κάνουν μαζικές παρακολουθήσεις. Γιατί να το κάνουμε αυτό χωρίς κανένα λόγο. Γιατί ο σκοπός αυτής της μαζικής παρακολούθησης και της διεύρυνσης δεν έχει καθοριστεί καθόλου. Δεν θα πρέπει, συμφωνώ, με αυτό που είπε ο κ. Μπόνια, δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα όσα λέει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα συνεργαστώ μαζί σα, θα υποβάλω τροπολογίε, αλλά μόνο για να ενισχύσουν περαιτέρω την πρότασή σα. Γιατί συμφωνώ απόλυτα με την κατεύθυνση που έχετε πάρει. Ευχαριστώ. Η κυρία Έρνστ από την Γκουε. Μάλιστα. Και εγώ σκεφτόμουν και άκουσα τις παρεμβάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε με σαφήνεια ότι εδώ πρόκειται για ένα μέσο για την ενίσχυση της ασφάλειας και του απόρριτου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Πρόκειται για ένα βασικό εργαλείο. Χαίρομαι που η συγκήτρια με τέτοιο καλό τρόπο πρότεινε τα ζητήματα αυτά. Το σχέδιο πραγματικά είναι πολύ καλό και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε την περαιτέρω δουλειά. Και επίση ε, πιστεύουμε ότι φυσικά η εναρμόνιση με τον GPDR και με τον κανονισμό για την ε, ιδιωτική σφαίρα θα πρέπει να είναι κάτι το δεδομένο. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ναι, εδώ θα επιμείνω. Και ακολουθώ την λογική των προτάσεων. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για δύο άρθρα. Για το άρθρο 8 Εδώ είναι σημαντικό το ότι διευκρινίζεται ότι οι χρήστε δεν μπορεί να του αρνηθούμε την ε, πρόσβαση αν δεν συνεννούν σε επεξεργασία των δεδομένων που δεν είναι απαραίτητη. Αυτό είναι σαφές, δεν διατυπωθεί με τον τρόπο αυτό και το ζητήσαμε και στο GPDR. Και είναι σημαντικό να υπάρξει διευκρίνηση. και τα θέματα της συνένεσης ε, για την σύναψη της ε, σύμβασης. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι πολύ απλό να το κατανοήσουμε, αλλά να κατανοήσουμε ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Το 2 β η διαγραφή αυτού, όπου μιλάμε για το χρήστη. Η λύση που προτείνει η συγγητρία και στην τροπολογία 89 και 90. Δεν ξέρω κατά πόσον, κατά πόσον επιλύει το γρίφο. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο και ίσως καταθέσουμε δική μας πρόταση. Το άρθρο 11, το ότι δεν έχουμε διαπιστώσει ιδιαίτερο ενθουσιασμό, δεν νομίζω ότι προκαλεί εκπλήξη σε κανέναν για την αποθήκευση των δεδομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα το ε, καταπολεμούσαμε, αλλά είναι καλό που στο άρθρο 11 ε, επισαρχόμαστε λίγο στην ουσία της ε, προβληματικής και στο άρθρο 23.2 του GPDR αναφέρεται. Το υποστηρίζουμε αυτό σε κάθε περίπτωση και θα πρέπει να σκεφτούμε στη τελική ανάλυση ποιο θα είναι το τελικό προϊόν. Αν εφαρμόζεται δηλαδή το άρθρο το, όπως το προτείνει η Ευρωπαϊκή η Συγκεντρία. Μετά από... Ε, θα έχουμε 28 ξεχωριστούς εθνικούς νόμους για την αποθήκευση. Αυτό το κομμάτι από τα άρθρα 11 θα πρέπει να αφαιρεθεί, πιστεύω, προκειμένου τουλάχιστον εδώ να υπάρχει ευρωπαϊκή και μόνο αρμοδιότητα. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι για μένα. Για την τεχνική οδητηρότητα, το είπε ο κ. Μπόνι, το υποστηρίζουμε κι εμεί θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή ή φιλικότητα προς το χρήστη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και τονίζουμε χωρίς ε, καμία αμφιβολία. Αυτά στην παρούσα φάση και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την ε, εισηγητρία σας. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριο από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε και φυσικά όλοι γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα είναι φιλόδοξο και είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τις τροπολογίες. Χαίρομαι που έχουμε χρόνο μέχρι τις 10 Ιουλίου. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα καταφέρετε μέχρι τότε. Και προσβλέπω ιδιαίτερως και στις διαπραγματεύσεις με την εισηγήτρια και όλους τους κοιόδης. Επιτρέψτε μου ένα-δύο σχόλια γενική φύσεως. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και πάλι ότι πρόκειται μια διάταξη, για μια διάταξη λέξη σπεσιάλη στο GPDR. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ισχύει το GPDR στις πιο πολλές περιπτώσεις και μόνο πραγματικά εάν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη για τον κανονισμό ή privacy θα πρέπει να υπάρξει τέτοια ε, εξειδίκευση των διατάξεων όπως προβλέπεται στο κείμενο του GPDR. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ενδεχομένω να είναι πραγματικά σημαντικό να υπάρξουν περαιτέρω διευκρινήσεις στον κανονισμό για το θέμα του πότε εξειδικεύεται ο GPDR και αν χρειάζεται να υπάρξει αναφορά στο GPDR σε κάθε περίπτωση ή αν ισχύει γενικά και δεν χρειάζεται να υπάρχει διευκρίνηση κάθε φορά. Εδώ κάπως θεωρώ ότι όλοι δεν κατανοούμε από ακριβώς ποια είναι η νομική σύνδεση εγώ θα είχα την εντύπωση ότι θα έχει νόημα πραγματικά σε πρώτη φάση, σε πρώιμη φάση, να ζητηθεί από την νομική υπηρεσία να διευκρινίσει λίγο αυτή τη σχέση λέξη σπεσιάλης μεταξύ GPDR και του κανονισμού για το e-privacy, για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί έχω την εντύπωση ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι 100% λογική σε ό,τι αφορά τη σχέση αυτή ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα ήταν ε, πραγματικά χρήσιμο να έχουμε λίγο παραπάνω γνωμοσύνη και λίγο παραπάνω ενημέρωση για το τι γίνεται. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρθηκα, στο οποίο αναφέρθηκα και στην πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων. Πιστεύω ότι ο πολιτικός πώς θα πρέπει να είναι σαφές και προς τα έξω, ότι δεν μειώνουμε τα εφιστάμενα δικαίωματα των Ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών σε ό,τι αφορά την προστασία του στο διαδίκτυο. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Και αυτό γιατί βλέπουμε όλο και πιο πολύ ότι υπάρχει tracking και στο διαδίκτυο και με στα τηλέφωνα, στο ίντερνετ των πραγμάτων, ακόμα και τα αυτοκίνητά τους, ακόμα και τα ρούχα τους ενδεχομένω να τους ε, παρακολουθούν και να τους καταγράφουν, τα καταστήματα από τα οποία περνάνε. Οι πόρτε των καταστημάτων. Όλο και πιο πολύ tracking, όλο και πιο πολύ παρακολούθηση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το δικαιολογήσουμε σε όλους ε, τους α, ε, ε, μα ότι σε αυτές τις συνθήκες μειώνουμε την προστασία. Και σε διάφορα αφορά το GPDR θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε ως γενική προσέγγιση. Όλα τα υπόλοιπα ασφαλώς υπόκεινται στην κατανα... κατανοήση του πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα δικαιώματα, πώς μπορούμε να χρεώσουμε τις ε, επιχειρήσεις να εφαρμόζουν όλες αυτές τις προδιαγραφές. Για παράδειγμα, με θέματα συνένεσης. Πώς δίβεται η συνένεση. Είναι σωστή ιδέα να γίνεται αυτό μέσω των ρυθμίσεων του browser. Μήπως υπάρχει καλύτερη λύση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ καλύτερη λύση από αυτό που κάνουμε τώρα με τα cookie banners. Αν κάποιος έχει καλύτερη ιδέα, ας τη συζητήσουμε. Αυτή την προσέγγιση θα ήθελα να ακολουθήσουμε, να βρούμε την καλύτερη λύση σε κάθε περίπτωση. Τέλος, μία πρόταση, επιτρέψτε μου να κάνω, μία παρατηρήση να κάνω για την καταμέτρηση Εγώ πιστεύω ότι στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να κινηθούμε προ την κατεύθυνση τη συνένεση. Αν γινόταν αυτό στον αναλογικό κόσμο, όπου για παράδειγμα εγώ μπαίνω σε ένα κατάστημα και ξέρω τον ε, ιδιοκτήτη του καταστήματο. και αυτό ενδεχομένω να φτιάχνει το προφίλ μου, να μαζεύει πληροφορίε για μένα, για να μου δώσει καλύτερα προϊόντα στο μέλλον, για να μπορεί να στοχεύσει καλύτερα σε μένα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό επιτρέπεται, γιατί αυτή τη σχέση δεν ξεκινά από τη στιγμή που μπαίνω στο κατάστημα. δεν θέλω, να μπαίνω στο κατάστημα καν. Αν υπάρχουν άλλοι 40 άνθρωποι όμως μέσα στο κατάστημα, εγώ αυτό που θέλω είναι αυτοί οι 40 πελάτες να είναι πραγματικοί πελάτες, να μην με παρακολουθούν και να με παρακολουθούν να θα πάω και στο επόμενο κατάστημα. Αλλά αυτό ακριβώ συμβαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στο website τα οποία δεν τα ξέρω. Δεν τα έχω ξαναδεί στη ζωή μου και δεν ναι, με παρακολουθούν μόνο στο συγκεκριμένο κατάσταση. Με παρακολουθούν και στο σπίτι μου, με παρακολουθούν και στο επόμενο κατάστημα, στο αυτοκίνητό μου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε, το επιθυμούμε. ή ε, τουλάχιστον να ξέρω ότι θα με ρωτήσουν μία φορά αν ε, συμβαίνει αυτό. Ιδάλλως θα χάσουμε διάφορες αξίες που έχουμε θέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω στη συνεργασία με τους Κιώδης. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πέτρος. Και τώρα να ακούσουμε και τα μέλη τη Επιτροπή ο κ. ο οποίο είναι ε, ο εισηγητή από πλευρά τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να αναρωτηθούμε τι θέλουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ψηφιακή αγορά και να προωθήσουμε τον τρόπο αυτό την ευρωπαϊκή οικονομία, την ελεύθερη ροή δεδομένων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάπως, αν είναι δυνατό. Και τα βασικά μα ε, δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ό,τι αφορά τα άρθρα 7 και 8, επίσης να τα υποστηρίξουμε. Αυτό όμως που παράγουμε στην Επιτροπή είναι ότι ξεκινάμε με την αρχή αυτή και τελικά καταλήγουμε να λέμε ότι όλα είναι επικίνδυνα και όλα ενδεχομένω να πλήξουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Δεν θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Και αυτό μου θυμίζει την ε, ιρανική θρησκεία που ξεχνάνε σε πολλές περιπτώσεις ότι ο κόσμος γύρω τους αλλάζει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα έπρεπε να κάτσουμε και να κοιτάξουμε λίγο πιο έντονα μήπως μπορούμε να πετύχουμε μια καλύτερη ισορροπία από αυτή που έχουμε ως τώρα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι ήταν ήδη οπισθοδρομική. Δεν έχουμε κατά νου ότι υπάρχει το GPDR το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση όλων αυτών. Και τώρα συνεχίζουμε λοιπόν στο ίδιο πνεύμα. Η έκθεση της συναδέλφου. Λάουριστιν. Θεωρώ ότι όντως ε, δεν ε, έχει την συνεκτικότητα που θα επιθυμούσαμε. Καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε γιατί χρειαζόμαστε μάλλον λέξεις σπεσιάλες, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι το GPDR αποτελεί τη βάση. Και υπάρχουν και επιπλέον και κάποιοι άλλοι κανόνες οι οποίοι έχουν να κάνουν με το απόρριτο της επικοινωνίας. Συνεχίζουμε. Και ακόμα και η επικέντρωση του να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο σύστημα για τη συνένεση δεν θεωρώ ότι προωθεί τη νομική βεβαιότητα. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί τα ίδια δεδομένα δεν υπάρχουν στο ίδιο, στην ίδια νομοθεσία. Τα μεταδεδομένα, τα μεταδεδομένα όπως αποτελούν ενδεχομένω μια νέα κατηγορία δεδομένων. Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος. Πρόκειται για τη τελική ανάλυση για προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει να υπάγονται στο Γενικό Κανονισμό για τα προστασία των προσωπικών δεδομένων και στι σχετικέ αντιτάξει. Η επικέντρωση σε θέματα συνένεση θεωρώ ότι είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, γιατί η συνένεση οδηγεί σε κατάργηση της ιδιωτικής ζωής όλο και πιο πολύ. Και γι' αυτό λοιπόν το ότι επικεντρωνόμαστε σε αυτή τη συνένεση θεωρώ ότι αποτελεί λάθος ε, τρόπο και θα πρέπει να το διαπιστώσουμε αυτό. Τουλάχιστον να καταργήσουμε το λέξη specialis και κατά δεύτερον να δημιουργήσουμε απόλυτη α, συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για να αποφύγουμε τη σύγχυση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, θα μπορούσε να, τι προβλήματα θα μπορούσε να σημαίνει μια τέτοια λύση. Και τέλο, δεν καταλαβαίνω. Στην τροπολογία 13, για παράδειγμα, λέμε ότι χρειαζόμαστε συνένεση, αλλά για περαιτέρω επεξεργασία θέλουμε νέα συνένεση. Εδώ σύμφωνα απόλυτα με τον συνάδελφο Ντάλτον. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διάκριση από το άτομο σε ό,τι αφορά αυτές τις πολλαπλές επεξεργασίες τελικά καταλήγουμε να εκνευριζόμαστε με τη συνένεση και κάποια στιγμή θα σταματήσουμε να διαβάζουμε το τι συνενούμε. Αυτό πιστεύω ότι είναι λάθος λύση. Και γιατί λοιπόν το direct marketing ρυθμίζεται με τέτοιο μη ικανοποιητικό τρόπο. Μη ικανοποιητικό θεωρώ εγώ. Θεωρώ ότι στο οικονομικό σύστημά μας θα πρέπει να έχουμε λύσεις opt-out, ένστασης. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, αλλά γιατί είμαστε τόσο περιοριστικοί στην προκειμένη περίπτωση. Δεν το κατανοώ. Για τα cookies. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή των cookies, αλλά στις τροπολογίες ξεπερνάμε και τον GPDR. Η τροπολογία 83 για παράδειγμα, τι εννοεί. Ότι θα επιτρέπονται και cookies τρίτων μερών. Στο άρθρο 10 θα έλεγα για την συμπλήρωση του GPDR. Το άρθρο 8 τροποποιείται σημαντικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει για τη διαγραφή των δεδομένων στο σημείο αυτό. Ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό και τη διάθεση των ε, κατευθυντηρίων γραμμών για τις ε, αρχές 119-121 τροπολογίε. Ε, τροπολογίες. Ήδη υπάρχει υπερβολικά πολύ γραφειοκρατία στα θέματα αυτά, είτε πρόκειται για την οδηγία, για τον κανονισμό, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά οδηγούν σε μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος. Το χρειαζόμαστε πραγματικά λοιπόν αυτό και κοιτώντας την τροπολογία υπαριθμών 110 θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαφωνιά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αν μου επιτρέψετε να τα σχολιάσω. Κοιτώντα την επικοινωνία α, μηχανήματος προς μηχάνημα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη συνένεση. μιλάμε για συνένεση από άτομα. Αυτό δεν αφορά τα μηχανήματα. Δεν είναι προετοιμασμένο το νομικό μας σύστημα για κάτι τέτοιο. Στην πρόταση 4, στην, στο άρθρο 4 της πρότασης υπάρχει μια αναφορά στον κώδικα επικοινωνίας. Θεωρώ ότι και η πρόταση για το e-privacy δεν μπορεί να ισχύσει τον κώδικα Επικοινωνία απαραίτητα. Γι' αυτό λοιπόν κατανοώντας την ιδέα ότι όλα θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, παράλληλα χρονικά, θεωρώ ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει νομικά. Γιατί οι επιχειρήσει πιστεύω ότι θα χρειαστούν πολύ πιο πολύ χρόνο για να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, σφάλμα μου, διότι είχαν ε, πολλά να πούν όλοι οι σκιώδεις, αλλά έχουμε τώρα πια πολύ λίγο χρόνο και Λυπούμε που έχει τόσο λίγο χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μιλήσει, διότι έπρεπε να έχω σταματήσει νωρίτερα τους άλλους συναδέλφους, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση στις 12 για να ψηφίσουμε κιόλας μετά. Ε, πέντε λεπτά λοιπόν και μετά θα επανέλθει η Μαριού Λάουριστιν. Πέντε λεπτά γιατί υπήρχαν πολλά σημεία φιλεγόμενα από ό,τι ακούσατε. Και μετά ε, κάντε λίγη υπομονή γιατί ε, αφού ακούσουμε τα πέντε λεπτά της Επιτροπής και τη Μαριού Λάουριστιν, θα έχουμε τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ ευχαριστούμε που μας δώσατε λίγο περισσότερο χρόνο. Θα τον ε, χρησιμοποιήσουμε, αλλά θα δώσουμε χρόνο και στην κυρία Λάουριστην. Ευχαριστώ όλους και για την παρουσίασή τους και για τα σχόλιά τους, διότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ποικιλία απόψε εδώ. Κάποια από όσα υπόθηκαν για να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε τη συλλογιστική και τα αίτια για τα οποία προτείναμε ότι προτείναμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα για τους ορισμούς. Πολύ ε, καλό να ακούσουμε τις διευκρινήσεις της κυρίας Λάουριστην, διότι πραγματικά η δική μας ήταν να υπάρχει ευθυγράμμιση με τους ορισμούς του κώδικα και θα δούμε ότι θα συμφωνηθεί και εκεί στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας ώστε να έχουμε συνέπεια σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Κάτι που επανέρχεται διαρκώς στη σημερινή συζήτηση είναι η σχέση του GDPR και του e Είπε και ο κύριος Άλμπρεχτ ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια. Όμω είπε και η κυρία Λάουριστην ότι πρέπει να προσέξουν τα διαφορετικά πεδία. Εδώ μιλάμε για εμπιστευτικότητα επικοινωνιών. Επ' αυτού πολλά ακούστηκαν. Για τι επιχειρήσει λόγου χάρη. Γιατί καλύπτουμε και τα νομικά πρόσωπα και όχι μόνο τα φυσικά. Έτη, συσκευή προ συσκευή. Επικοινωνία. Όταν μιλάμε για εμπιστευτικότητα και απόρριτο, και αυτή είναι η διαφορά με το GDPR, έχει να κάνει με το τι συμβαίνει τη στιγμή τη εκπομπή τη επικοινωνία ε, για, για το απόρριτο όλων των επικοινωνιών. Εάν δεν καλύψουμε τα νομικά πρόσωπα, όταν μια μικρή επιχείρηση επικοινωνεί με μια άλλη, δεν θα καλύπτεται. Δεν καλύπτεται από το GDPR, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Είναι πολύ σημαντική η αγορά ε, και το μέτρο έχει αυτό στο ε, μυαλό τη. Και ε, επιτρέπουμε έτσι να λειτουργήσουν καλύτερα online οι επιχειρήσει. Επίση, οι συσκευέ ε, ε, όταν λειτουργούν απομονωμένα, εφόσον αποστέλουν δεδομένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά να σκεφτούμε το παράδειγμα τη ηλεκτρονική υγεία, έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα όπου η αποστολή δεδομένων και τα ηλεκτρονικά δεδομένα της υγείας δεν καλύπτονται από το GDPR. Αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε εδώ. Θα είναι επικοινωνία συσκευή προς συσκευή. Πρόκειται λοιπόν για άλλη μια περίπτωση, για τα browser. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην επιβάλλουμε default ρύθμιση, να απαιτούμε πληροφόρηση και ο καταναλωτής να κάνει την επιλογή. Ο κύριος Μπόνι ανέφερε ότι Πρέπει στην αγορά να υπάρχει περιθώριο ώστε ε, η τεχνολογία να βρει τη λύση για τον τελικό χρήστη. Τώρα, γιατί πρέπει να επενθυμίζουμε στους χρήστες, αυτό που είπε και ο κ. Ντάλτον, γιατί πρέπει να επενθυμίζουμε στους χρήστες την επιλογή τους. Βάσει του εμπορικού, του δικαίου του εμπορικού δικαίου πρέπει να θυμίζονται στους καταναλωτές ε, οι σημαντικές επιλογές που έχουν να κάνουν. Δεν, τα περισσότερα κράτη θα κάνουν αυτό. Δεν θα ήταν λοιπόν ε, περίεργο να ήταν πιο ε, αυστηρή η νομοθεσία των εμπορικών συναλλαγών και του δικαίου των καταναλωτών από ότι το e-privacy θα είχαμε ένα πρόβλημα εδώ. Γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε περισσότερη διαφάνεια απλώς. Τώρα για, τα, για τις ρυθμίσεις των browser νομίζω το κάλυψα και Παραμένουμε στη διάθεσή σας. Απλώς να σας θυμίσω γιατί χθε είδαμε να δημοσιεύεται από τη Eurostat μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για την ασφάλεια των πληροφοριών. Και εκεί είδαμε την χρήση των δεδομένων που βάσει της μελέτης αντικτύπου μας μπορούμε να μην επιτρέπουμε τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημίσεις. 40% των Ευρωπαίων καταναλωτών έχουν περιορίσει τη δράση τους ε, στα κοινωνικά δίκτυα ε, για να αποφύγουν τους, ε, τη χρήση των δεδομένων για σκοπούς κατανάλωσης και εμπορικούς. Ευχαριστώ να ήταν χρήσιμο όσο είπα και παραμένουμε στη διάθεσή σα για τη συνέχεια τη διαδικασία με το πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Για το χρονοδιάγραμμα να πούμε ότι νομίζουμε ότι πολύ καλά θα συμβαδίσει αυτό που έχετε προγραμματίσει με τον GDPR και την εξέλιξη της έκθεσης. Αυτό είχε προτείνει αρχικά στο χρονοδιάγραμμα και ο κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ του συναδέλφου που συμπίεσαν τι ε, παρεμβάσει στο τέλο, αλλά είναι σημαντικό για ένα τέτοιο νομοθετικό φάκελο να προλάβουμε. Συνάδελφοι, να έχουμε πρώτα και την ε, συγκίτρια και μετά να περάσουμε στις προφορίες. Um, <clears throat> uh, uh, Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης εισηγητές, τον κύριο Φως, φυσικά την Επιτροπή για τη συζήτηση αυτή. Είμαι ευγνώμων για κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που κάνατε. Φερρυπίν, θα πρέπει να στραφούμε αμέσως προς το νομική υπηρεσία για να μας κάνει αυτή τη διευκρίνηση σε ό,τι αφορά τον κανονισμό προστασίας των δεδομένων και την, το e-privacy ε, ως ε, λέξη specialis που πρότεινε ο κύριος Άλμπερτ. Ε, καλό θα είναι η απάντηση να δοθεί πριν από το, μάλλον το φθινόπωρο, όταν ξεκινήσουμε. Τώρα για τα συγκεκριμένα προβλήματα που εντόπισαν οι σκιώδεις εισηγητές, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ εκτενείς συζητήσεις για όλα αυτά τα προβλήματα και θέλω να πω μόνο το προφανές για την προσέγγιση Ντάλτον. Προφανώς κύριε Ντάλτον έχουμε πολιτικές διαφορές ε, αλλιώς καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει η ιδιωτική σφαίρα των προσώπων εμείς και αλλιώς εσείς. Και χαίρομαι με αυτά που είπατε κύριε Φως, γιατί χαίρομαι που σε αυτή την Επιτροπή δεν λέμε πρώτα οι επιχειρήσεις και μετά τα δικαιώματα των προσώπων. Όχι σε καμία περίπτωση μια τέτοια προσέγγιση θα περάσει εδώ. Προς, προσβλέπω λοιπόν σε μια εντατική συνεργασία. Χαίρομαι με την προθεσμία που θεσπίσαμε και τέλος να ευχαριστήσω και τον και τις υπηρεσίες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ήμασταν σε συνεχή επαφή. Σας είπα ήδη από την αρχή ότι ήταν ε, τόσο συνεχής ε, και αδιάσπαστη αυτή η συνεργασία που έχουμε την αίσθηση ότι δεν ε, σταμάτησε ποτέ. Ευχαριστούμε Μάριον για την πολύ σκληρή δουλειά που κάνεις και τους κοιόδους ηγητές επίσης για τη συνεργασία. Το πολύ σκληρό χρονικό διάστημα 10 Ιουλίου είναι η προθεσμία ε, για την υποβολή των τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του, θα ψηφίσουμε μάλλον τον Οκτώβριο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε δύο, σε δύο λεπτά, συνάδελφοι, για τις ψηφοφορίες. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε όταν όλοι ετοιμαστείτε με τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες αναχείρας. Okay, everyone in place? Καθίσατε όλοι, πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Με το σημείο 7. Ψηφίζουμε για την έκθεση για τα ασοφωνιστικά συστήματα και συνθήκες. Η κυρία Μπέργκισον θέλει να πάρει το λόγο σύντομα. Όχι, συγγνώμη, η συγκήτρια. Σας ευχαριστώ για την ψηφοφορία. Ένα κοινό κείμενο γιατί οι σκιώδεις συζητητέ ε, με υποστήριξαν πάρα πολύ και σε τεχνικό και σε ηθικό επίπεδο και τους ευχαριστώ για την σύνταξη του κειμένου. Πολλοί μίλησαν για μεταφραστικά προβλήματα. Ήθελαν η τελική μετάφραση για το κείμενο να στην, που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια να είναι πολύ ακριβής, ειδικά σε ό,τι αφορά τους νομικούς όρους η κυρία Κινίτσι, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει τον, ή μάλλον ανησυχεί για τον όρο regime, καθεστώς, γιατί δεν είναι ακριβώς ε, ο ίδιος στα αγγλικά και στα, στα γαλλικά, μάλλον και στα ιταλικά. Και ένας τσέχος συνάδελφος ανησυχεί για τη μετάφραση κάποιων λέξεων. Και εγώ είμαι νομικός και ανησυχώ για διάφορους, ε, διάφορους όρους, όπως παραδείγματος χάρη η τα δικαιώματα δημιουργού, droit d'auteur στα γαλλικά, που μεταφράζεται copyright. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Copyright είναι το αντίθετο από το ε, δικαιώματα δημιουργού. Σας ευχαριστώ και καλή ψηφοφορία. Ευχαριστούμε κυρία Μπερζερόν. Παρακαλώ καθίστε και βάλτε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες στη σχισμή. Ξεκινάμε το συμβιβασμό 9. Ψηφίζουμε. closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 22. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 19α. Ψηφίζουμε τώρα. Συγγνώμη, ε, λέει ο επίδειξα τον συμβασμό 12. Θα ψηφίσουμε τώρα τη συμβαστική τροπολογία 12. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρα προφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19α. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7α. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική τροπολογία 15. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. και τροπολογία 110. Πέρας. Τροπολογία 110, επαναλαμβάνω. Ψηφίστε ακόμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110. Πέρας πέρα Πέρας ψηφοφορίας. Συγγνώμη, 111. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 112. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρόεδρε. Μπορώ να ψηφίσω διανατάσσεως χειρός γιατί ξέχασα την κάρτα μου. Μπορώ. Φυσικά δεν μπορώ να σας πω όχι. Προφανώς μπορείτε. Εντάξει. Τι θα κάνουμε. Να σηκώνετε αντίχειρα για το ναι ε, το, προς τα κάτω για το όχι, τα κλασικά βέβαια και θα σας ε, καταμετρούμε και εσάς. Θα σας προσθέτουμε. Συμβασμός, συμβαστική τροπολογία 19. Πες, Εγκρίνεται. Τροπολογία 126. Πέρας. Απορρίπτεται. 127. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε, τροπολογία 130. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απορρίπτεται. 133. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12α. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 149. Πέρας. Εγκρίνεται. 150. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Πέρας. Εγκρίνεται. 155. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 156. Πέρας. Εγκρίνεται. 157. Πέρας. Υπορρίπτεται. 158. Πέρας. Εγκρίνεται. 159. Πέρας. Εγκρίνεται. 173. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός υπέρφων 11. Πέρας. Εγκρίνεται. 182. Τροπολογία 182. Πέρας. Εγκρίνεται. 186. Πέρας. το κολλαγή 187. Πέρας. υπορρίπτεται. Τροπολογία 201. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 220. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 247. Πέρας. Συμβαστική τροπολογία 21. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 264. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 265. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 267. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 268. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 269. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 270. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 272. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 281. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 283. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές. Ψηφίζουμε μαδικά. Πέραν από τις α, τροπολογίες 90 και 19. Ψηφίζουμε λοιπόν τι αιτιολογικές αναφορές on block. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. απορρίπεται συγγνώμη. Απορρίφθηκε. 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Επίσης απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. 20. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται το ψηφοριό Πέρας. Απορρίπτω. 37. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 3. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται του ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 56 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. 57 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Συμβαστική 7. άρχη του ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, η 76. Άρχη του ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρχη του ψηφοφορία. Πέρας. 88 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 92 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 94 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται με 44 ψήφους υπέρ, 4 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Κυρία Μπεχζεγού, σας συγχαίρουμε. Κλείσαμε και με τις προφορίες και λίγη και συνεδρίαση για σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ.